Uh, Καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τη συνεδρίαση. Προσοχή παρακαλώ. Conversations. Thank you. Σταματήστε τη συζήτηση παρακαλώ. was yesterday. Το σημείο 21. Αντιπροσωπή στην Κύπρο. το συζητήσαμε χτες. Έχετε μία, ένα έντυπο στο φάκελό σας. Μικρή η αντιπροσωπεία, λιγάριθμη, τριμελής, ο υποφαινόμενος Πίτερ Στνάσνη και ο Ιωάννης Κασουλίδης που ήρθε. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές επισκέψεις στην Κύπρο. Μας δίνουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ανταλλάξουμε απόψεις με την κυβέρνηση, αλλά και με βουλευτές, με ενδιαφερομένους κύκλους εδώ με το εμπορικό επιμελητήριο, με τα συνδικάτα και επιτόπου να σφιγγομετρήσουμε τα συναισθήματα του κόσμου για την Προεδρία. Πρώτη Προεδρία ενός νέου πρόσφατου μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσης, της Κύπρου, μιας μικρής χώρας και είναι μια δυνατότητα να δούμε επιτόπου και το σειρματόπλεγμα και τη διαχωριστική γραμμή εντός της Λευκοσίας, της πρωτεύουσα της Κύπρου. Αυτό επιβεβαιώνει ότι είναι χρησιμότατες οι επισκέψεις και αισθάνομαι ότι ενισχύεται τη θέση μου να τεθεί τέρμα σε αυτού του είδους επισκέψεις. Απ' την άλλη, αν δεν κάνουμε αυτές τις επισκέψεις, τι μας απομένει στην Ένωση για να κάνουμε επισκέψεις εμείς σαν Επιτροπή. Υπάρχουν σχόλια μήπως. Ουχή. Ας μπούμε λοιπόν στην σημερινή μέρη σε διάταξη, σημείο 22. Τροπολογία κανονισμού του Συμβουλίου για το dumping. Είναι δεύτερη τροποποίηση του κανονισμού λόγω αποφάσεως του δικαστηρίου όχι του πάνελ διαθετήσεως διαφορών του ΠΟΕ αλλά του δικού μας του δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού μήνα Φεβρουάριο λοιπόν το ΔΕΚ αποφάσισε ότι οι τεχνικές δειγματοληψίες που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον καθορισμό της αντιμετώπισης τη οικονομία αγοράς δεν συμμορφώνονται με τον βασικό κανονισμό και τις ρυθμίσεις αντι-dumping. Οπότε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να εισαχθούν διατάξεις στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διευκρινίζουν τις διαδικασίες έρευνας, το πώς αποφασίζονται οι δασμοί για παραγωγούς εκτός των δειγμάτων και να μην υπάρχουν χρονικά όρια για να, υπάρχει, για να καθοριστεί κατά πόσο η αγορά αντιμετωπίζεται με τους κανόνες ελεύθερης αγοράς. Αυτά περί του κανονισμού, εγώ είμαι εισηγητής. πρότασή μου είναι να ακολουθήσουμε με απλουστευμένη διαδικασία. Υπάρχουν οι σχετικοί κανόνες του Κοινοβουλίου επ' αυτού και λέω να υιοθετήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άνευ τροποποίησεως και οι συντονιστές συμφωνούν. Αν συμφωνείτε θα λάβει η χώρα σήμερα η ψηφοφορία. Και όλα αυτά για επιτάχυνση της διαδικασίας. Ας ξεκινήσει η συζήτηση. Πολ Μέρφυ, ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνω, χρειάζεται δειγματοληψία και ίσως δημιουργηθεί μεγάλο διοικητικό άχθος αν δεν αλλάξουμε κάτι. Η τροποποίηση του άρθρου 2.7 C λατινικό είναι πολύ σοβαρή δεν υπάρχει κανένα χρονικό όριο. Το τρίμηνο έφυγε και δεν αντικαθίσταται από 4, 5, 6 μήνε. Αντικαθίσταται, μάλλον διαγράφεται. Και αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό για του παραγωγού και τις μη ε, που θεωρούνται ότι δεν συμμορφώνονται με την οικονομία τη αγορά. Και γιατί, ποια είναι η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα ευρύτερο χρονικό όριο, αντί να καταργείται εντελώ, να μην υπάρχει κανένα χρονικό όριο που προβλέπεται. Άλλα σχόλια, παρατήρηση. Είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο πρόεδρο Θα τους ακούσουμε, λέει. Φαμπρίτσιο Νταπρίλε. Έχει το λόγο. Διευκρινήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ναι, ίσω θα πρέπει να πάω κατευθείαν στο ερώτημα που ετέθη για την RCT τη τρίμηνη προθεσμία για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίε κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση στου κανόνε τη ελεύθερη αγορά. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι προτείνει να αρθεί αδίποτε προθεσμία για να γίνει αυτό ο καθορισμό. Γιατί έχουμε διπλό λόγο. Πρώτον, η πρόσφατη απόφαση του ΔΕΚ διατείνεται ότι η παράταση της προθεσμίας είναι λόγος κατα καταργήσεως του τέλους του ε, αντι και αυτός είναι σοβαρός νομικός κίνδυνος. Και από την εμπειρία μας, όσον αφορά έρευνες για την οικονομία της αγοράς, έχουν δείξει ότι γίνεται περιπλοκότατο και χρονοβόρο ζήτημα αυτό. Το να λέμε ότι δεν υπάρχει καμία προθεσμία, κανένα χρονικό όριο δεν απολύτω ορθό, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει προσωρινά ε, τον ένα το μήνα της έρευνας όπου όλα τα απορίσματα για την καθορισμό της αξίας και αυτό αφορά και την συμμόρφωση με την οικονομία της αγοράς, περιθώριο dumping, ζημίες κλπ. κατά των συμφερόντων της Ένωσης πρέπει να γίνουν όλες αυτές, ε, αυτοί οι υπολογισμοί. Η διαγραφή της ενδιάμεσης προθεσμίας για την έρευνα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτός ο καθορισμός γίνεται το αργότερο στον ένατο μήνα της έρευνας, μαζί με τα άλλα απορίσματα της έρευνας. Ε, δεν θεωρούμε ότι αυτό ε, ότι είναι σοβαρό ή ότι είναι ένα είδος ποινής, αν θέλετε, επιβαρυντικό, διότι δίνει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα θεσμικά όργανα να καταλήξουν σε μια σωστή απόφαση εμπεριστατωμένη όσον αφορά την όλη κατάσταση για τις εταιρείες που λειτουργούν σε ματεβατικές οικονομίες. Άρα αυξάνεται κατά κάποιο τρόπο η ποιότητα και η λεπτομέρεια της έρευνας σχετικά με αυτό και γι' αυτό ε, κάνουμε αυτή την πρόταση. Διαφορετικά θα έλεγα ότι η πρόταση πράγματι είναι εστιασμένη τροπολογία αλλαγή ε, όσον αφορά το βασικό κανονισμό κατά του ντάμπινγκ, οπότε μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιεί για την οικονομία τη αγορά, τι μεθόδου δειγματοληψία για την έρευνα για συμμόρφωση με του κανόνε ελεύθερη αγοράς και αυτό ευθυγραμμίζεται πλήρω με τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής ε, σύμφωνα με τον ΠΟΕ και αυτό ο φορέας ε, διαθέσει των διαφορών του ΠΟΕ σε έκθεσή του το ανέφερε όσον αφορά τα τέλη αντιτόμπινγκ για τα υποδήματα. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια, λέει ο Πρόεδρος. Ουχή. Οπότε, προχωρούμε. Κοινή συζητήσει για τα θέματα 23 και 24. Ο Πάμπλο Σάλβα είναι ο εισηγητής και για τα δύο θέματα. Σχετίζονται με τη συμφωνία που δημιουργεί Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και της χωρών της Κεντρικής Αμερικής από την άλλη. Μία από τις εκθέσεις είναι προσωρινή για όπου άπτεται τη ΣΑΦΕΤ και άλλη έκθεση αφορά τη σύσταση για τη σύμφωνη γνώμη για την, αυτή τη σύνθετη ε, διεθνή συμφωνία. Είναι μια πλήρης εμπορική συμφωνία. Συζητήθηκε ήδη το θέμα. Ας γίνει δελεχέστερη συζήτηση όμως. Υπάρχουν τα σχέδια εκθέσεων. Υιοθέτησε χθε θέση το Συμβούλιο. Πρόχτες, 10 Ιουλίου, απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεπώς, έχει επιληφθεί για σύμφωνη γνώμη. Πιθανότατα αυτή θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Υπάρχει και σχετική διαδικασία για την πρόταση κανονισμού με μεταδιαφύλαξης. Ήθιστε αυτό στις εμπορικές συμφωνίες για το μηχανισμό σταθεροποίησης για τις μπανάνες Δεν σε εμπορικέ συμφωνίε, αλλά σε συμφωνίε με χώρε Κεντρική Αμερική είναι. Ο κ. Λάιχτριγκ είναι ο ε, Θα ψηφιστεί σήμερα η έκθεση. Draft reports. Λοιπόν, είπαμε σε 1, 23 και 24 θα συζητήσουμε. Θα δώσουμε το λόγο στον Πάμπλο για να μιλήσει και για τις δύο συμφωνίες. Έχεις το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω εσάς και να ευχαριστήσω και όλη τη γραμματεία η οποία βοήθησε για αυτή την έκθεση. Ε, είχαμε επίσης ε, αυτή τον ε, ανταγωνισμό σχετικά αφορά τις αρμοδιότητες και τελικά μπόρεσε να, να βρει την διέξοδο η γραμματεία. Η Επιτροπή μας επομένω, ήταν πάρα πολύ δραστήρια όσον αφορά αυτή την ε, εμπορική συμφωνία με την Κεντρική Αμερική της 29ης έκτου στη Γουαθικάλπα. Επίσης την ε, Τρίτη, όπως είπε και ο Πρόεδρος, το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση ούτως ώστε να κάνουμε αυτή την ε, απόφαση την απόφαση αυτή ε, και πρόκειται αυτό να επισημοποιηθεί ούτω ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να την επικυρώσει στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Σήμερα δε έχουμε ε, το άρθρο 50 το οποίο ρυθμίζει την ε, συνθήκη αυτή και την επικύρωση της. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει η έγκριση δηλαδή, την Επιτροπή μας στις 18 Σεπτεμβρίου και έτσι θα μπορέσουμε να επιψηφίσουμε την ε, σύσταση όσον αφορά αυτο τον τριμερή διάλογο στις 11 ε, Οκτωβρίου. Πρόκειται επομένως τώρα για πάρα πολύ σημαντική συμφωνία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την Κεντρική Αμερική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρόκειται επομένως ε, για ε, ε, κάτι το οποίο ισχύει από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες περιοχές του κόσμου και είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια η Κεντρική Αμερική και επομένως ε, ελπίζουμε ότι θα γίνουν και άλλες ε, τέτοιες συμφωνίες στο μέλλον, ούτω ώστε να έχουμε μια πολιτική ολοκλήρωση στην Κεντρική Αμερική, μια που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Επομένω, και, και ο Παναμά μας επομένως είναι σημαντική χώρα. Τώρα όσον αφορά την εμπορική πολιτική πρόκειται για μια ευκαιρία και για εμά και για την άλλη πλευρά, ακόμα για ένα βήμα επομένω ε, για αυτή την ε, πορεία που άρχισε το 1984 με τον διάλογο του Σαν Χωσέ και κορυφώνεται τώρα με αυτή την συμφωνία. Τώρα επομένως θα έχουμε επενδύσεις, θα έχουμε εμπορικέ ροές, θα έχουμε πολυμέρεια και επίσης θα έχουμε περισσότερη κοινωνική συνοχή με αυτό το ευρύ νομικό πλαίσιο που θα παρέχει ασφάλεια και έτσι θα έχουμε βαθμία απελευθέρωση των συναλλαγών, των υπηρεσιών, των ε, δημοσίων συμβάσεων στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Και ε, αυτή τη συνεργασία πρόκειται να διευκολυνθεί η προσαρμογή της Κεντρικής Αμερικής στις προκλήσεις αυτού του συμφώνου και θα συμμετάσχουν περισσότερο της Κεντρικής Αμερικής στη, στο, Διεθνή Φόρα και η Διεθνής Ένωμη Τάξη έτσι από πλευράς ε, εργασιακής και κοινωνικής ε, τώρα πρόκειται να ισχύσει με αυτή την συμφωνία σύμφωνα με τα όσα ε, έχει προβλέψει ο ΠΟΕ. Αυτό θα αφορά και τις γεωγραφικές ενδείξεις, τα φυτογειονομικά, τα περιβαλλοντικά. Πρόκειται επομένω για φιλόδοξο στόχο για ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα και έτσι όμω θα έχουμε περιφερειακή ολοκλήρωση όπως προείπα και θα έχουμε περισσότερη κοινωνική συνοχή ε, με τη βάση των αρχών του κράτους δικαίου και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται για την συνεργασία, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για το εμπόριο. Και έτσι επιβεβαιώνονται οι οι ε, στόχοι διεθνούς πολιτικής και, και των δύο πλευρών. Έχουμε μόνος τώρα πάρα πολύ στενούς, ε, πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς και θα τους ενδυναμώσουμε και επομένως τώρα θα είναι ε, πιο εύκολες οι ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, βιώσιμη ανάπτυξη και των δύο πλευρών και επομένως τώρα θα έχουμε τα θεμέλια για καλύτερη σχέσεις και των πλευρών του οπότε Τώρα θα μια νέα όθηση στις σχέσεις μας και επομένως ελπίζω συνενετικά να επιψηφίσουμε αυτή την συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να τηρήσει τα συμπεφωνημένα μόλις η συμφωνία αυτή τεθεί σε ισχύ. Παύλος, ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Συζήτηση τώρα. Ξεκινούμε βεβαίω πάντα με τους σκιοδησηγητές, ο κ. Λάχτφιντα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και κύριε εισηγητά. Πάρα πολύ σωστή ήταν η συνεργασία μας για το θέμα. Και επίσης, νομίζω ήταν ε, υπέροχο τα όσα έκανε η γραμματεία. Δεν νομίζω ότι θα τα είχαμε καταφέρει αλλιώς. Συμφωνώ με όλα όσα είπε ο εισηγητής. Και δεν ήθελα να τονίσω κάποια σημεία. Ε, τώρα το θέμα είναι το πόσο επηρέασε το έργο μας η Επιτροπή Εξωτερικών. Βέβαια. Δεν νομίζω ότι ήταν όρθο ε, από νομικής πλευράς το ότι αποφασίσαμε να ανοίξουμε την πόρτα στην Επιτροπή Εξωτερικών και στο πόσο επηρέασε τα πράγματα νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει αυτή η επιρροή της μιας επιτροπής του έργο της άλλης. Τόσο μας αφορά κάποια άλλα νομικά προβλήματα, τα πήγαμε καλά και όσον αφορά το περιεχόμενο, τέτοιε εμπορικέ συμφωνίε. δεν είναι μόνο εμπορικέ. Αφορούν θέματα πολλά πέραν του εμπορίου. Το Κοινοβούλιο νομίζω με επιτυχία χειρίζεται αυτό το, τη διασύνδεση εμπορικών θεμάτων με τα άλλα. Με τα άλλα όπως το περιβάλλον, όπως την εργατική πολιτική. Εδώ νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε τις χώρες με την εμπορική ισχύ μας. Νομίζω ότι αυτό με την εν λόγω συμφωνία το πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής με αυτόν τον τρόπο και σας ευχαριστώ. Well, you are quite right about competence. Uh, ναι, έχετε δίκιο όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Ναι, θα έπρεπε το να δική μας αρμοδιότητα. Αλλά δεν το σκέφτηκαν έτσι αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία. Τέλος πάντων. Τώρα, Μαρία, στο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση την οποία στηρίζω και θέλω να κάνω μία σκέψη. Ε, ελέγχθη προηγουμένως για τις επιτροπές αλλά έχω και ένα δεύτερο σχόλιο. Αυτή η συμφωνία εμπορικά είναι εξαιρετική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω καμία αμφιβολία επ' αυτού για τις ε, εταιρείε υπηρεσιών, για τις ε, χρηματικές χρηματοοικονομικές ε, επιχειρήσεις ε, και θα ανοίξει νέους ορίζοντας. Ελπίζω όμως ότι δεν θα ξεχνάμε και θα συμφωνήσουν ελπίζω οι συνάδελφοι ότι η συμφωνία δεν πρέπει μόνο να είναι προς όφελός μας αλλά και υπέρ της ε, βιώσιμης ανάπτυξης της Νοτιού Αμερικής και της ανάπτυξης του ε, τοπικού ε, κοινωνικού ιστού της βελτιώσεως των συνθηκών εργασίας δηλαδή μια συμφωνία συνδέσεως για μας δεν πρέπει να είναι απλώς ένας τρόπος να αυξήσουμε τις ε, ελεύθερες συναλλαγές αλλά θα πρέπει να αποβλέπει και στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των εργαζομένων ε, στην ε, Λατινική Αμερική για την προώθηση ε, της βιώσιμης ανάπτυξης, την προστασία των πρώτων υλών να μην αμφισβητηθούν, πρόσβαση στο, στο νερό και αυτό δεν πρέπει να αμφισβητείται και ελπίζω ότι ο συνάδελφος θα λάβει υπόψη όλες αυτές τις παρατηρήσεις και να είναι συμμετρικά προς όφελος η συμφωνία αυτή όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και των πολιτών που ζουν εκεί. Τώρα ε, η κυρία Κέλλερ εν ονόματι των Πρασίνων. Συμφωνώ με αυτά που ελέγχθησαν για τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως για τους εταίρους μας αυτή τη συμφωνία και στα πλαίσια αυτά έχω ορισμένες αμφιβολίες εάν η συμφωνία είναι προς όφελος όλων, διότι υπεγράφει την 30 ε, ε, επέτειο του παραξικοπήματος στην Ονδούρα και αν μιλάμε ε, για κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν πρέπει να παραβλέπουμε ένα τόσο σημαντικό γεγονός όπως το πραξικόπημα στην Ονδούρα. Δεν ξέρω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει αυτό το γεγονός, αν έχει κάτι να σχολιάσει επ' αυτού και όσον αφορά αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν ε, νομίζουμε ότι ε, διατυπώνεται εκπαρκώς στη συμφωνία ή ε, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και θα ήθελα να γνωρίζω εάν οι συμφωνίες αυτές συνάδουν με τις οδηγίες για την υποδομή της αγοράς στην Ευρώπη. Μπορείτε να μας το σχολιάσετε. Επιπλέον ξέρετε ότι κατακρίνει ο Σάι και άλλοι και είναι το βασικό σημείο της, του ξεπλήματος βρωμικού χρήματος από ε, την ε, διακίνηση ναρκωτικών όπως την Κολομβία. Μπορείτε να μας πείτε πώς όλα αυτά θα επηρεάσουν τις εξελίξεις ή εσείς αν έχετε λάβει υπόψη σας όλα αυτά τα γεγονότα. Όσον αφορά την ε, συμφωνία συνεργασίας που είχε συνάψει η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003 και η οποία ποτέ δεν εφαρμόστηκε από ό,τι ξέρουμε. Άλλαξε κάτι. Υπάρχει πάντοτε το ίδιο καθεστώς και αν δεν έχει αλλάξει κάτι ε, μπορείτε ε, να μας πείτε ε, τι έχετε κάνει για το PCA που έπρεπε να έχει ληφθεί η υπόψη για την ανάπτυξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη που ε, και τα σχόλια που υπάρχουν από αυτού εις ε, τη συμφωνία αυτή δεν είναι πολύ επικοδομητικά και πιστεύω ότι αποτελούν μια σημαντική αδυναμία διότι για μας ε, μια τέτοια συμφωνία συνδέσεως δεν θα προωθήσει ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε και την ανάπτυξη και δεν θα εξασφαλίσει κάλυψη αναγκών των χωρών με τις οποίες συναλλασσόμαστε. Ε, για την ΚΟΕ, ποιος ε, είναι εκπρόσωπος εδώ, ο Πολ Μέρφι. Νομίζω ότι η συμφωνία αυτή είναι τυπική των συμφωνιών που προσπαθεί να συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τον κόσμο που ενδιαφέρονται ιδίως για το ελεύθερο εμπόριο και ε, να προωθήσουν τις μεγάλες, ε, τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων της Ευρώπης παραβλέποντας τα συμφέροντα του, των λαών και ε, ε γι' αυτό τα στολίζει κανείς και με λίγα λόγια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχε καταλήξει ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει ισοτιμία με τη Συμφωνία της Κεντρικής Αμερικής ενώ η κατάσταση έχει χειροτερέψει και ιδίω όσον αφορά την βιοπικιλότητα και την διατροφική ασφάλεια. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να αντιταχθείτε σε αυτές τις εξελίξεις και ε, ποια είναι η κοινοβουλευτική διάσταση διότι βλέπουμε ότι και στο ΑΣΕΝ δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, οπότε τι θα κάνετε για να προωθήσετε ε, ε, το κοινοβουλευτικό πλαίσιο. Αφού κανείς άλλος δεν έχει σχόλια θα ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, βλέπω ότι έχουμε ε, τον κύριο Ματίας Γιούργενσεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Τζον Κλάρκ. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Εσείς είστε της Γενικής Διευθύνσεως ε, εμπορίου και ξεκινάτε, ο κύριος Γιούργενσεν. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Καταρχήν, συμφωνώ πλήρως με το γεγονός ότι πρόκειται για μία φιλόδοξη πρόταση που πρέπει να χαιρετήσουμε που είναι προς και των δύο περιοχών και διευκρινήθηκε στις διάφορες μελέτες των ε, ε, ε, του αντικτύπου των επιπτώσεων ε, που έχουν γίνει ε, είτε από το Κοινοβούλιο είτε από την ε, Επιτροπή και προσπαθούμε να υπάρξει μία περιφερειακή ε, ολοκλήρωση ε, οικονομική και εμπορική στην περιοχή και έχουμε και ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλω να τονίσω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη πολιτική προσήλωση των χωρών ε, της Κεντρικής Αμερικής και χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή του εις της ακροάσης που οργάνωσε η Επιτροπή ΙΝΤΑ και στην υπογραφή στις 29 Ιουνίου στην Κεντρική Αμερική και οι έξι πρόεδροι των χωρών της Κεντρικής Αμερικής παρίσταντο στην υπογραφή με τους υπουργούς εξωτερικών και τους υπουργούς εμπορίων που υπέγραψαν τις συμφωνίες με τον Επίτροπο Κάλντε Γκούχτ και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τώρα θα θέλαμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην διαδικασία κυρώσεως στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Κεντρική Αμερική κατά τρόπον ώστε και οι δύο πλευρές να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία η οποία ε, έχει διαπραγματευτεί και ολοκληρωθεί προδιετίας. Όσον αφορά τα, τα βασικά σχόλια τα οποία έθεσαν ορισμένοι ευρωβουλευτές, καταρχήν ε, υπάρχει ένα βασικό και ισχυρό κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης στη συμφωνία, υπάρχουν νομικοί, και δεσμεύσει για τις χώρες οι οποίες πρέπει να εφαρμόσουν ε, οικολογικές πρακτικές στην αλληλεία ε, ε, και δημοκρατικές διαδικασίες και υπάρχει και μία διαδικασία εποπτείας από ένα πάνελ κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες αυτές θα σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και αυτό θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική ε, συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην ενίσχυση της δημοκρατίας στην Κεντρική Αμερική. Τίθεται και ένα άλλο ερώτημα. Ε, ο Παναμάς και η Κωνσταντίνα Ορισμένοι δηλαδή ε, βουλευτές έχουν θέσει το ερώτημα αυτό εάν ασχολούμαστε παρκώς με, και αν εξετάσαμε το εάν ο Παναμάς και η Κωνσταντίκα είναι φορολογική παράδειση τι κάνουμε επ' αυτού και καθ' όλες τις ε, διαπραγματεύσεις εμείς είχαμε θέσει το θέμα με τις εμπλεκόμενες χώρες της Κεντρικής Αμερικής και στη συμφωνία έχουμε περιλάβει ε, δύο ε, άρθρα, το ένα που αναφέρονται στην ε, χρηστή διακυβέρνηση και στο πολιτικό και στον οικονομικό τομέα και τα τελευταία χρόνια ο Παναμάς και η Κωνσταντίνα έχουν προσχωρήσει σε 12 συμβάσεις και στα πλαίσια του ΟΣΑ και όλες ε, αυτές οι χώρες προσπαθούν να προσαρμόσουν την νομοθεσία τους στη διεθνή πρότυπα κατά τρόπον ώστε να ε, διαγραφούν από τον αρνητικό κατάλογο του ΟΣΑ όσον αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος νομίζω και τη δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί από αυτού αντιλαμβάνομαι ότι είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι πρέπει κανείς να διατηρήσει την δυνατότητα να ε, ε, υπάρξουν οι προϋποθέσεις και η νομοθεσία για την για την προώθηση των οικονομικών υπηρεσιών οι δε χώρες αυτές θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλήματος δρόμικου χρήματος. Βέβαια θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή σας επί του βασικού αυτού φακέλου και ελπίζω ότι θα υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Ο κύριος Τζον Κλάρκ. Για τις μπανάνες έτσι, για τη γεωργία αν θα είναι υποφελής η συμφωνία για τις μικρές ε, εκμεταλλεύσεις, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις σε κάποια εταιρική περιοχή. Η συμφωνία προβλέπει ευρύτατη πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόντα όπως ρούμι, ζάχαρη, μπανάνες, τροπικά φρούτα, ξηρούς καρπούς, βόλιο κρέας. Βελτιώνεται για όλα τα προϊόντα η πρόσβαση και αν δείτε τη σύνθεση του αγροτικού τομέα στην περιοχή. Δεν είναι όλα πολυεθνικά, δεν είναι λατιφούντια όλα. Ε, υπάρχει μεγάλη ποικιλία μικρών εκμεταλλεύσεων οικογενειακών και δεν χρειάζεται να υποθέσει κανείς ότι δεν ωφελούνται όλοι οι γεωργοί από τη συμφωνία. Θεωρούμε ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι μικρές εκμεταλλεύσεις θα ωφεληθούν από την πρόσβαση στην αγορά που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μας τη συμφωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, να πω κάτι για αυτό που είπε ο κύριος ε, Πολ Μόρφη για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή που προβλέπεται από αυτή τη συμφωνία. Είναι σαφές για μένα και πρέπει να ξεκάθαρο για την Επιτροπή το εξής ότι αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα έχει δικαίωμα εποπτείας της συμφωνίας και εφόσον η συμφωνία έχει και πυλώνα εξωτερικής πολιτικής και εμπορικό, ε, αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να υπάρχει όσον αφορά την εποπτεία της εφαρμογής ε, του τρίτου πυλώνα της συμφωνίας. Και θέλω αυτή η Επιτροπή να είναι πολύ ε, στεναρή, κυρίως όσον αφορά την καταπολέμηση για το ρόλο μας σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή. Ευχαριστώ Πορ Μέρφη που το θέσατε αυτό το θέμα και θα έπρεπε να είναι σαφές από την ε, αρχή. Ο Πάμπλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όσα σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Λάιτφριτ, ευχαριστώ τον κύριο Λάιτφριτ για την συνεργασία του. Νομίζω ότι ήταν πάρα έξοχη ομάδα που σχηματίσαμε. Χαρά μου που συνεργάστηκα μαζί σα. Συμφωνώ με τον κύριο Λάιχτφριντ. Ε, συμφωνώ με τη θέση του όσον αφορά την ε, πολύ μεγάλη επιρροή της Επιτροπής ΑΦΕΤ και δέχτηκα την πρόταση να μειωθεί αυτή η επιρροή υπερβολική στο μέλλον. Όσον αφορά τα σχόλιά του για το περιεχόμενο της έκθεσης, συμφωνώ ότι τα εμπορικά και μη εμπορικά θέματα πρέπει να συνδέονται, συμφωνώ μαζί σας, αλλά πάντα επικοδομητικά. Όσα αυτά που είπε η κυρία Σαρνέθ, Συμφωνώ. Κυρία. 100% συγκεκριμένα αυτά είπατε όσον αφορά την εμπορική συμφωνία. Είναι νομίζω τέλεια, υπέροχη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Και τώρα η πρόκληση είναι το πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε, πώς θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε την βιώσιμη ανάπτυξη τη Κεντρική Αμερική. Γιατί για άλλη μια φορά σα λέω ότι ελπίζω ότι με αυτή τη συμφωνία θα βοηθήσουμε την ε, πολυμορφία, την οικονομική τη Κεντρική Αμερική, την κοινωνική συνοχή τη Κεντρική Αμερική και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Και κατά αυτόν τον τρόπο, επίση, νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερη αμοιβαιότητα σε επίπεδο κοινωνικό και περιβαλλοντικό τώρα όσον αφορά αυτά τα οποία είπε η κυρία Κέλεφ. Επίση επίσης και ε, με εκείνη συμφωνώ όσον αφορά το πραξικόπημα δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι κάτι το οποίο στην ε, Ονδούρα ε, ξεπεραστεί και γι' αυτό και πιστεύω ότι με αυτή τη συμφωνία ε, θα βοηθήσουμε την κατάσταση ούτως ώστε στο μέλλον μην έχουμε τέτοια γεγονότα ε, και ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ε, επανάληψη φαινομένων και καθ' αυτόν τον τρόπο νομίζω θα θωρακίσουμε τη δημοκρατία της περιοχής της χώρας τώρα στον Αποδίκη ε, δεν συμφωνώ σε σχέση με, το, με τις θετικές συνέπειες για την Κεντρική Αμερική αυτές τις συμφωνίες γιατί νομίζω ότι έτσι νομίζω ότι θα έχουμε τα εργαλεία θα θα δώσουμε, θα δώσουμε κάποια μέσα, κάποια εργαλεία στις κυβερνήσεις και της Αμερικής τόσο ώστε να μπορέσουν να έχουν κάποιο είδους αγιαφόρο ανάπτυξη, ε, να βοηθήσουμε την οικονομία τους και κατά αυτόν τον τρόπο θα του βοηθήσουμε και να ε, του βοηθήσουμε να εκμεταλλευτούν αυτή τη συμφωνία και καμία αμφιβολία ότι αυτό πρόκειται να ωφελήσει την ε, κεντροαμερικανική οικονομία τους τώρα όσον αφορά την εποπτική επιτροπή Συμφωνώ, Πρόεδρε. Όλοι, όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Χωρίς καμία επιφύλαξη πρόκειται να συμφωνήσουμε και νομίζω ότι αυτή η Υποπτική Επιτροπή πρόκειται να έχει πάρα πολύ σημαντική, σημαντικό ρόλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, απλώς επαναλαμβάνω σε όλους τους ευχαριστίες μου. περιμένουμε πώς και πώς το θα γίνει η προσωρινή θέση και του συμφώνου προθεσμία για τις τροπολογίες για την προσωρινή έκθεση. 19 του μηνός το μεσημέρι τροπολογία για, τη, για την διαδικασία σύμφωνης γνώμης στις 20 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία το μεσημέρι. Χτες μας ενημέρωσαν και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας είπαν ότι συμφωνούν να εφαρμοστούν οι εφαρμοστικές διατάξεις από την απόσταση του Συμβουλίου και αυτές οι διατάξεις προσθεθούν στον κανονισμό με τον διαφύλαξης της Συμφωνίας Σύνδεσης με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Πάμε το επόμενο σημείο είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία, πρέπει να περιμένουμε ένα πεντάλεπτο. Μικρή διακοπή πέντε λεπτών. President, shall we start? Okay, voting. Πολύ ωραία, πρόεδρος και τώρα ήρθε των ψηφοριών. Well, before we... Πριν να αρχίσουμε την ψηφορία, Λέει ο πρόεδρος, επιτρέψτε να σας πω ότι έχουμε κάποια νέα μέλη της Επιτροπής μας. Οπότε με μεγάλη μου χαρά. Καλώς ορίσατε κυρία Νοραμπέρα. Καλώς ορίσατε. Αντικαθιστάτε ε, τον κύριο Μπάτ. Και τον Χένρι Βέμπερ. Αν θα αντικαταστήσει τον κύριο Αρίφ. Θα του πω και με τα καλωσορίσματα όταν τον δω. Η Επιτροπή μας. Με μεγάλη μας χαρά σας, καλωσορίζουμε για το σώστον να ε, μοιραστείτε μαζί μας τόσα ενδιαφέροντα κάνουμε. The first uh, item to be voted is item Το πρώτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι το υπαριθμό 25. Το 25 είναι. Εφαρμόγη τη διμερού ρήτρα διασφάλιση και του μηχανισμού σταθεροποίηση για τι μπανάνε στο πλαίσιο τη Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεντρική Αμερική. Um, we have 20, ε, 65 amendments. Amendment 9. 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική. Υπαριθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, λέει, αυτό ήταν το πρώτο τμήμα. Έχουμε κατά διέρεση ψηφοφορία. Δεύτερο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 3 υπέρ. Κατά. Υπέρ. Κατά. Αποκλείσει. Το δεύτερο τμήμα. Τι είναι υπέρ. Κατά. Αποκλείσει. Εγκρίνεται, θα ηλεκτρονικό έλεγχο. ψηφίζουμε. ψηφίζουμε. Ένας σοσιαλιστής παραπάνω. Πέρας ψηφορίας. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. Δώδεκα. Γεωργίε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Υπέρ ξαναλέω πρόεδρος. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε ηλεκτρονικά έλεγχο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. 20. Against Thomas And the vote is closed. And it was not correct. Rejected. απορρίπτεται, δεν επιψηφίστηκε. Ah, yes. My, my eyesight is not as good as... Ah, Α, αυτό το ότι δεν, δεν είμαι αυτός που ήμουνα, δεν βλέπω το ίδιο καλά. Α, τελικά όχι, 16-12. Εγκρίνεται, εγκρίνεται τελικά. Σαράντα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Γεωργίας, 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε. Για να δούμε. Γεωργίας 13. Ψηφίζουμε. The vote is closed. And it was rejected. Α, τελικά απορρίφθηκε, λέει ο Πρόεδρος. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Τροπολογία υπαριθμών 21. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23. Και μαζί Γεωργίας 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται Γεωργίες 10 5 καταπίπτει 45 υπέρ 25 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Γεωργίες 16 Γεωργίας 16. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Εγκρίνεται. Γεωργίας. Γεωργίας 18 και μαζί τροπολογία 27 του εισηγητού. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γεωργίας 20 και 29 υπέρ κατά εγκρίνεται. Γεωργίας 2 υπέρ κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την υπερθμόν 2 Γεωργίας. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Πού είμαστε? Μόνο ένα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθυμών 2. Κατά διαίρεση. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα της ε, ιδίας τροπολογίας. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. Γεωργία, υπαριθμών 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 6. Υπέρ. γεωργίας Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρισμόν 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα, Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε, Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι, Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Γεωργίες, οκτώ Υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται Επτά, υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Γεωργίας 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική υπερθυμών 6 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γεωργίες. Παριθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και η τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. επί της προτάσεως της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 25-1. Δύο εποχές. Το σχέδιο του νομοθετικού ψηφίσματος τώρα ψηφίζουμε. Πέρας. το ίδιο αποτέλεσμα. 25, 1 με δύο εποχές. Συγχαρητήρια προς τον ε, εισηγητή κύριο Λάχτριτ. Είκοσι τώρα. Εφαρμογή τη διμερού ρήτρα διασφάλιση και του μηχανισμού σταθεροποίηση για τι μπανάνε στο πλαίσιο Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκή Ένωση. Κολομβίας και του Περού. Ο κ. Λάγκεν είναι ο εισηγητής. Και έχουμε εδώ τι υποστάσεις αυτές τροπολογίες του εισηγητού και 15 από άλλους βουλευτές. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία υπαριθμών 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 2. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 3. Κατά διάρρηση. Πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Συνδυαστική, Παρακτημόν 3, Ξεφύγουμε. Πέρας. Δεκατέσσερα. Ηρεμία, ηρεμία παρακαλώ. 14 υπέρ κατά αποχέ. Α, απορρίπτεται. 15 υπέρ. Ψηφίζουμε. Το 14. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Γεωργίας. 12. Υπέρ. Κατά. Δεν κρίνεται. Έλεγχος για την 12 Γεωργίας. Ψηφίζουμε. Απορρίπτωτα. 16. Υπέρ. Κατά 17 υπέρ. Πώς? 16. Επιμένετε. Well, you have the right. Uh, ναι, ναι. Δικαίωμά σα. Έλεγχο επομένω για το 16 ψηφίζουμε. 16 ψηφίζουμε. <laughs> Amendment Amendment 17 17 in favor 17 υπέρ κατά να απορρίπτεται Check Amendment 17 Έλεγχος ηλεκτρονικός για το 17 ψηφίζουμε πέρας Όντω απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Παχέ εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 13 Γεωργία. 18 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπερθυμών 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 20 και 14 γεωργίες, συμβαστική 5, υπέρ καταποχής εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 8, υπέρ κατά εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 23 και Γεωργίας 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γεωργίας 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ιτιολογικές παράγραφοι Γεωργίες. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα και τρία Γεωργίες. εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα γεωργίε υπέρ κατά Αποχές. Α, απορρίπτεται. Τέσσερα, γεωργίες. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. μόνο τρία. Πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Γεωργίας. Έξι συμβαστική υπέρ κατά πέρα της ψηφοφορίας. Ε, τροπολογία. Γεωργίας υπερθυμών. 6 κατά υπέρ αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπερθυμών 6 εις δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, πέρα, κατά. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Πέντε, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Έξι, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Γεωργίες, επτά, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Οκτώ, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Γεωργίας 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περθμόν 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γεωργίας 9 υπέρ. Γεωργίας 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γεωργίας ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τέλος η η 24 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε για το 24. Ναι, απορριφθήκε. Τελική ψηφοφορία ψήφισμα την πρώτη επιτροπή όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Μια ψήφο κατά και τρεις απόχέ. Τώρα, ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματο. Ψηφίζουμε. Πέρας. το αποτέλεσμα είναι το ίδιο 26, 1 χωρίς αποχές, συγχαρητήρια εισηγητά. Well, regarding the, the two files that have voted on, regarding the... Σε σχέση τώρα με τη, τα δύο αυτά θέματα και την συμφωνία σύνδεση με την Κεντρική Αμερική, δεν έχω κάποιο αίτημα σε σχέση με τις πρώιμες διαπραγματεύσεις σε αυτή τη φάση. Εγώ πρώτα θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια και ο ίδιος ο συγητής, ο Λάχτφιντ, μας είπε ότι δεν θα ήθελε να ζητηθεί εντολή όσον αφορά με το Συμβούλιο. Και συμφωνώ μαζί σα Σίγητα, όπως πάντα. «27 τώρα. Θέμα 27. Σε σχέση με τον κανονισμό περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου εξαγωγών μεταφοράς μεσητείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης. Φιέλνερ. Ψηφίζουμε. Εκεί ψηφοφορίας. Τέσσερα υπέρ, κατά. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παριθμόν 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5-5 για το 5 έλεγχος. 5. Πέρα τις εφορίες. Amendment 9. That's your right. Το είναι 9. Ναι, ναι, ναι, δικαίωμά σας. 9, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, έλεγχος, ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. δέσμη τροπολογιών. υπάρχουν ένα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Για τη δέσμη 1. Δέσμη υπαριθμών ένα. Πέρας. Απορρίπτεται. Παριθμόν 2. Περ, κατά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτη δέσμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. Τελογικές παράγραφοι Παραθμόν. Ε, ναι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την πρόταση επιτροπής όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 14-5 με 10 αποχές. Προχωρούμε τώρα στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Ψηφίζουμε. Πέρας. 15. 4. 10. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια εισηγητά. Κύριε Φιόλνας. Έχει ζητήσει σύντομη δήλωση ο Σίγητας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την έκθεση για τη Ρωσία, θέλω να πω σε το ξέρουν ότι η Ντούμα έκανε μια οριακή ψηφορία χθε το πρωί και ψήφισαν υπέρ της προσχώρησης εις τον ΠΟΕ. Η Επιτροπή μας θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. But before... Πρόεδρος. Πριν ταξιδέψουμε στη Ρωσία, έχω να σας πω, όσον αφορά την τελευταία ψηφοφορία, ότι ο εισηγητής προτείνει να αρχίσουν επίσημες διαπραγματεύσεις με Συμβούλιο και Επιτροπή για συμφωνία σε πρώτη αναγνώση από τη βάση της εντολής για την δημοτευτική ομάδα όπου θα συμμετάσχει ο πρόεδρος, ο εισηγητής και οι σκιώδες εισηγητές. Και όπως γνωρίζετε, εγώ Είμαι κατά οποιασδήποτε πρώιμης συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Βεβαίω μπορεί να ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Για να δούμε ποιο συμφωνεί με την πρόταση του εισηγητού. Ψηφίζουμε. Όχι, όχι, όχι για τη Ρωσία. Πρόκειται για την έκθεση Φιόλνερ. Πρόκειται για πρόταση για μια πρώιμη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε αυτήν την έκθεση όλες οι ψηφοφορίες ήταν οριακές. Δεν υπήρξε σαφής πλειοψηφία. είχαμε ε, απόσχεια, αλλά αλλιώ θα την, ε, αν δεν είχαμε την αποχή, θα την είχαμε απορρίψει. Όμω προτείνω να πάμε στην Ολομέλεια και μετά να κάνουμε πούμε για τι διαπραγματεύσει. Το να πάμε διαπραγματεύσει πριν την Ολομέλεια δεν έχει νόημα, Πρόεδρο. Να σα πω τι γίνεται, γιατί κατά κανόνα εγώ είμαι κατά οποιασδήποτε πρώιμη συμφωνία από την ιδίω όταν έχουμε ευρωπαϊκή ψηφοφορία στην Επιτροπή. Διότι οι πολιτικέ ομάδε δικαιούνται να συζητήσουν τις απόψεις ή στην Ολομέλη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος για μια προηγουμένη συμφωνία ή πρώτη ανάγνωση, γιατί αυτό θα ε, παραβιάσει το δικαίωμα αυτό των πολιτικών ομάδων να συζητήσουν τις απόψεις και κατόπιν να υπάρχει μια διαπραγμα... εντολή διαπραγματευτική από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή μας. Οπότε αυτό το πρεσβεύω παγίως και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Και όταν υπάρχει εντολή από την Ολομέλεια, αυτό είναι ισχυρότερα εντολή. Οπότε οι κοινοβουλικέ ομάδε τότε δεν μπορούν να παραπονεθούν μια που έχουν εκθέσει και συζητήσει ή στην Ολομέλη. Επομένω, κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτό το οποίο ζήτησε ο εισηγητής. Θα πρέπει να τηρήσουμε την ε, αρχή μας όσον αφορά το θέμα. Κύριε Φιόνιλα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, συμπαθάτε μου για να ξεκαθαρίσουμε το εξή. Όχι, τι λέτε, δεν, δεν έχει μιλήσει ο εισηγητής. Δεν ζήτησε τίποτα τέτοιο ακόμα ο εισηγητής. Νομίζω ότι θα ήταν λογικό. Αν δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν θα υπήρχε λόγος να ξαναρχίσουμε να εξετάζουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Από την άλλη μεριά θέλω να σας πω ότι δύο τροπολογίες καταψηφίστηκαν και επομένως το πιο σωστό είναι να κάτσουμε και να δούμε τι προαγγίψε. Εγώ πάντως νομίζω ότι ακόμα και αν καταψηφίζατε θα, θα αποσπούσα εγώ την πλειοψηφία. Τέλος πάντων, είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε τόσο ισχυρή εντολή για διαπραγματεύσεις. Άρα, δεν είναι ιδιώδη τα πράγματα. Άρα, με κάποιο είδου ε, fast track διαδικασία να πάμε στην Ολομέλεια και α γίνει και εκεί μια. Δεν, δεν, δεν ανησυχώ ιδιαίτερο πρόεδρο. Καλά, τότε το αίτημα απεσύρθη. Σοφής απόφαση, Κρίστοφερ Φιόντα. Ευχαριστώ. Point uh, item 28 uh, about which uh, Robert Sturdy has... Σημείο 28. Ο Sturdy. Sturdy. important information. Εδώ σημαντικές ε, πληροφορίες μάλλον. Έχουμε 21 τροπολογίες. και οκτώ συμβαστικές λέει ο Πρόεδρος. Start with the compromise amendment. Συμβαστική υπαριθμόν 8. Υπέρ. Against abstentions. Carried. Υπέρ κατά εγκρίνεται τώρα η συμβαστική υπαριθμόν 1. Ε, Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται η συμβαστική υπαριθμόν 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. 11. Υπέρ. Κατά. Άσυγχρονα ήμουν αφηρημένος, έχετε δίκιο. 11. Έλεγχος. ψηφισμού. Πέραση ο Απορρίπτωται. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμών 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κατά αποχές 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο της νομοθετήσεως όπως τροποποιήθηκε ψηφίζουμε. And vote is closed. And it was carried by 26 votes in favor. Εγκρίνεται με 26, 3 και 1 εποχή. Συγχαρητήρια, κύριε Στέρντι, εισηγητά. Amendments uh, on the Council Regulation. Και τώρα λοιπόν το θέμα 29, που είναι τροποποίηση του κανονισμού για την άμυνα κατά των εισαγωγών dumping χωρών ε, τρίτων μη μελών. Σήμερα το πρωί αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την απλουστευμένη, απλοποιημένη διαδικασία. Δεν έχουμε τροπολογίες και ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 27 Μηδέν, δύο αποχές και προχωρούμε. Πακιστάν. Στο Πακιστάν, ναι, ναι. Χθες αποφασίσαμε για αυτή την ψηφορία. Να επικυρώσουμε, να συμφωνήσουμε με αυτήν την συμβαστική συμφωνία Κοινοβουλίου, Συμβουλίου. σας διενεμήθη και ψηφίζουμε. Τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται με 20, 0, 10 αποχες Δεν θα συγχαρώ τον εισηγητή λέει για τον εαυτό του πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία των ψηφοφοριών. Well Παρακαλώ καθίστε και όσοι αποχωρούν τις αιθούσεις σας το κάνουν ήσυχα. Και εκείνοι επίσης οι οποίοι έχουν αρχίσει την κουβεντούλα παρακαλώ να σταματήσουν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μείνουν στην αίθουσα. Παρακαλώ να ξαναρχίσουν την δουλειά. Έχουμε τώρα το θέμα. Υπάρχουν 21 ε, Μπορείτε. Με την η Ιαπωνία. Πρόκειται περί σχεδίου κειμένου. Sorry. Um, sorry, uh, there is the, still the item um, Ξεκολουθούμε να έχουμε τα 30, λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενώσης Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Τροφίμων. Είναι σχέδιο σύστασης, διεθνή συμφωνία. Αυτή είναι η διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Ήδη ε, το συζητήσαμε. Αναβεσβήτητα θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Στόχος η αύξηση προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στη Μολδαβία. Είμαι εισηγητής. Δεν έχω πρόβλημα να συστήσω στην Επιτροπή λοιπόν να συμφωνήσει με την ε, συμφωνία αυτή. Υπάρχουν σχόλια, παρατηρήσεις από την Ομίγυρη. Ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος είναι εδώ. Ο Τζον Κλάρκ έχει το λόγο. Δεν ήθελα το λόγο, ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς υποστηρίζει την αξιολόγησή σας και τα συμπεράσματά σας και ελπίζουμε η Επιτροπή να δώσει την σύμφωνη γνώμη της ε, τώρα σε αυτή τη συμφωνία. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 20 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Σημείο 31. Εμπορικές διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ιαπωνίας. Μου ζητήθηκε από την Ιαπωνική ραδιοτηλεόραση Japanese Broadcasting Company να μαγνητοσκοπήσει τις συζητήσεις για το θέμα αυτό. Δεν βλέπω γιατί να έχουμε αντίρρηση. Υπάρχει αντίρρηση. Οπότε τους δίνουμε την άδεια να μαγνητοσκοπήσουν. Όπως ξέρει το Κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούνιο ζήτησε από το Συμβούλιο να μην δώσει την έγκριση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων μέχρι να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της διαπραγματευτικής εντολής. Επανεπέμφθη το θέμα στην Επιτροπή μας και η Επιτροπή αυτή το εδώ συζητήσει. Σχέδιο πρώτας ψηφίσματος για την έναρξη διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. Ο μόνιμος συγγητής για η Ιαπωνία της Επιτροπής μας, επιφορτισμένος με το φάκελο, είναι ο Μάρτιν Κάζακ της Άρντε, στον οποίο δίνω παρευθύ στο λόγο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως προανεφέρθη, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε τον μήνα Ιούνιο ένα ψήφισμα και ζήτησε από το Συμβούλιο μη δώσει διαπραγματευτική εντολή για διαπραγματεύσει με την Ιαπωνία μέχρι να τοποθεθεί μέσω δεύτερου ψηφίσματος στο Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο ήδη διεξήγαγε ενδελεχή συζήτηση στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπορίου και το Σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εθετήσει σχέδιο οδηγιών διαπραγματευτικών στις 18 ε, Ιουλίου. Θα διαβεβαστεί το θέμα στο Συμβούλιο με έγκριση διαπραγματευτικής εντολής κάπου το φθινόπωρο. Οπότε έχουμε το σχέδιο ψηφίσματος, δεύτερου ψηφίσματος στους φακέλους, Βασίστε επί δύο αξώνων. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία βάσει των αποτελεσμάτων των βολιδοσκοπήσεων. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, να είμαστε προσεκτικοί στον αφορά διαπραγματεύσεις με ρήτες διαφύλαξης. Πιστεύω ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε τέτοιες συμφωνίες με μεγάλες οικονομίες το κάναμε με την Κεντρική Αμερική, Κολομβία και Περού. Αυτές οι συμφωνίες FTA Με αυτές τις χώρες καλές και άγιες ήταν, αλλά κλονίζεται η οικονομία μας και πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί στις διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί λοιπόν η ανάπτυξη να μόνο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το εμπόριο για να αναπτυχθεί η οικονομία μας. Δύο εταίρους έχουμε μπροστά μας. Η Ιαπωνία και η ΙΠΑ. Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο είναι η Ιαπωνία. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ήταν επιτυχείς στην Ιαπωνία είχαν τεράστια κέρδη. σε ένα σεμινάριο πριν από δύο μέρε είδαμε ότι η κατανάλωση η Ιαπωνική είναι δύο φορέ αυτή τη Κίνα. Τεράστιε δυνατότητε για την Ευρώπη. Όσο περιμένουμε δε, η Ιαπωνική συμμετοχή στην ε, εταιρική σχέση του ειρηνικού θα προχωρήσει. Πρέπει να κινηθούμε πριν τον ανταγωνισμό. Να κινηθούμε όχι αφελώς. Στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι δύσκολος τομέας. Χρειάζονται σκληρέ διαπραγματεύσει. Πρέπει να είμαστε αυστηροί όσον αφορά του όρου. Για να είναι υποφερή η μελλοντική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρω κάποιου όρου στην έκθεσή μου. Δεσμευτική ρήτρα αναθεώρηση πρώτα απ' όλα. Αν δεν υπάρχει πρόοδο όσον αφορά του χάρτε για προμήθειε κλπ. να ανασταλεί συμφωνία. Δεύτερον, πραγματικό άνοιγμα της Ιαπωνικής αγοράς, όχι θεωρητικό. MTB για τις προμήθειες που ξεπερνούν ε, τους οδικούς χάρτες. Πρέπει να υπάρχει δεσμευτικός μηχανισμός για να μην δημιουργηθούν νέα MTB. Οι ευρωπαϊκοί δασμοί θα πρέπει να έρθουν αν υπάρχουν επιτεύγματα όσον αφορά την Ιαπωνία. Ε, ε, μηχανισμός διαφύλαξης πρέπει να διαπνέει τη συμφωνία. Θέλουμε καλή συμφωνία για τις γεωγραφικέ ενδείξεις τις Ευρωπαϊκή και πρέπει να γίνει η δεύτερη αξιολόγηση συνεπειών μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ, να μην απαιτούμε υπερβολικά πράγματα. Η Ιαπωνία ήδη έχει κάνει υποχωρήσει, όπω ρυθμιστικέ αλλαγέ όσον αφορά τα βιολογικά τρόφιμα για του αερόσακου, για τα αυτοκίνητα και για δυνατότητα να εκδίδονται οι ε, διάφορες οδηγίες και τα διάφορα έγγραφα για τις κρατικές προμήθειες και στα αγγλικά. 30 προσανατολισμοί οδικοί χάρτες έχουν υιοθετηθεί για τα NDBs και ένα για κρατικές προμήθειες. Πόσα μπορούμε να ζητήσουμε πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Και το αίτημα για προκαταβολές είναι μια ε, δικαιολογία για να παρεμποδιστούν διαπραγματεύσεις. Αυτοί που δεν θέλουν διαπραγματεύσουν με την Ιαπωνία, τους ρωτώ, τι φοβόμαστε. Έχουμε εμπειρία άλλωστε στην Επιτροπή, με τη Μερκοσούρ, με την Άζεαν και το Συμβούλιο με τις χώρες του Συμβουλίου του Κόλπου. Και ξέρουμε ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθούν, πάση θυσία, όπως είπα στο σχέδιο ψηφίσματος, αν η Ιαπωνία δεν δείξει ότι είναι αρκετά φιλόδοξη, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διακόψει τι διαπραγματεύσει. Και αυτή είναι και η θέση του Επιτρόπου, από ό,τι είδα από τι συνομιλίε μαζί του. Επ' αυτού λοιπόν, πρόεδρε, συνάδελφοι, λέω ότι χρειάζεται αυτή η συμφωνία ελευθέρου μπορείου με, το, με την Ιαπωνία. Χρειαζόμαστε καλή συμφωνία και ελπίζω ότι τελικά να καταλήξουν σε καλή συμφωνία. Και ελπίζω και το κείμενο που ετοίμασα να μα βοηθήσει προ αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Μάρτιν. Όπως ξέρεις και εσύ, πριν από δύο μέρες, ο κ. Σοκάδα, υφυπουργό της Ιαπωνίας, ο αντιπρόεδρο τη κυβερνήσεω, είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο τη Ιαπωνίας αποφάσισε πολιτική για αριθμιστικές και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Θα ληφθούν αρκετά μέτρα που αφορούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε κατάλογο αποφάσεων που ελήφθησαν. Ας ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. ΕΛΚ. Κασπάρη. Έχεις το λόγο. Αξιόμενη κύριε Πρόεδρε, Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία, αλλά ε, έχω προβλήματα με αυτή την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, γιατί πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της ασκήσεως είναι ενδιαφέρον, αλλά όχι πολύ φιλόδοξο. Απ' την άλλη πλευρά γνωρίζω βέβαια ότι ε, είναι μία λογική προώθηση της συμφωνίας που υπογράψαμε για την ε, Κορέα και θα ήμουν πολύ ευγνώμων αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουμε θέσει και στην Ολομέλεια δηλαδή τι γίνεται με την Ταϊβάν που είναι στην ίδια περιοχή που σε πολλά, πολλούς τομείς πουλά και κατασκευάζει και πουλά παρεμφερεί προϊόντα και όπου υπάρχουν συμφωνίες. Εάν τώρα διαπραγματευτούμε με την ε, ε, Ιαπωνία θέλουμε σε δύσκολη θέση την Ταϊβάν ε, διότι θα έπρεπε να σκεφτούμε και τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων με άλλες χώρες της περιοχής για να μην βρεθούν χαμένες και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει το θέμα αυτό. Επίσης όσον αφορά την, ε, τον τίτλο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά αλλά πρέπει να σκεφτούμε και άλλες χώρες εκτός της Κορέας και της, ε, ε, της Νοτιού Κορέας και της Ιαπωνίας για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των λαών της περιοχής. Επίσης το θέμα της Ιαπωνίας για μένα διαφέρει από αυτό της Κορέας διότι αν δούμε ε, το, μέσο, το, το ποσοστό αγοράς που ε, είχαν πριν από τη ε, ε, ε, πριν από την σύναψη της συμφωνίας βλέπουμε ότι άλλαξε η αντιμετώπιση των Κορεατών και έκτοτε αυξάνουν τα προϊόντα που αγοράζουν και κατασκευάζονται εκτός Κορέας και πολλούνται εντός της χώρας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει αυτά που μας έχει πει, δηλαδή ότι αν δεν υπάρχουν πρόοδοι του ευρωπαϊκού εμπορίου προς την Κορέα που δεν έχουν σημειωθεί θα μπορέσει να υπάρξει μια επαναδιαπραγμάτευση διότι ε, εδώ μιλάμε για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου το σημειώνουμε έχουμε ε, κλείσει συμφωνία για το Περού, για την Κεντρική Αμερική. Έχουμε όμως πάρα πολλές συμφωνίες ε, ελευθέρου εμπορίου που δεν σημείωσαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια καμία πρόοδο και δεν είναι ούτε προς δικό μας συμφέρον ούτε των ε, ε, Ιαπώνων να ε, επεκτείνονται αυτές οι συμφωνίες και να μην υπάρχει καμία αναδιαπραγμάτευση. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσει ένα χρονοδιάγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει πόσο προσωπικό χρειάζεται και πόσο, πότε θα ξεκινήσουν οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Αλλά θα ήθελα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει την Ιαπωνία. Πρέπει να δούμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε εμείς να ανοίγουμε τις αγορές μας και οι Ιάπωνες να μην ε, δίνουν καμία ένδειξη ούτε ε, στα λόγια αλλά ούτε και στην πράξη ότι μπορούμε να προσχωρήσουμε στην αγορά τους διότι στο τέλος θα αντιμετωπίσουμε φοβερά προβλήματα. Ευχαριστώ κύριος Λάνιε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάζακ για το σχέδιο το οποίο παρουσίασε και πιστεύω ότι περιέχει πολύ σημαντικά στοιχεία διότι για μένα είναι αδιαφυσβήτητο ότι η Απωνία με την οποία έχουμε πάρα πολλές διαπραγματεύσεις κάθε χρόνο και ε, με την οποία ε, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες είναι ε, μας, πρόσχητες στα συμφέροντά μας και ως εκ τούτου είναι καλό να προσπαθούμε να έχουμε μία στενή συνεργασία και για πολιτικούς και για οικονομικούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει και ο κύριος Κάζακ το είπε αυτό σαφέστατα, Υπάρχει μία σειρά από μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια τα οποία δυσχεραίνουν την είσοδο στην εμπορική αγορά της Ιαπωνίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να συνάψουμε συμφωνίες θα πρέπει να απαιτήσουμε να εξαλειφθούν αυτά τα μη δασμολογικά εμπόρια και είναι πολλαπλά και πολύμορφα. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου θα υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Και θα παραθέσω εδώ τρία παραδείγματα. Όλοι οι εμπορικοί μας εταίροι έχουν ε, τις, ε, ε, έχουν υπογράψει τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου προβλέπεται η αμοιβαία αναγνώριση των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών τους. Μόνο η Ιαπωνία έχει εφαρμόσει ελάχιστο ενδιαφέρον και συμμόρφωση προς αυτόν τον κανονισμό και εδώ ε, λέγεται ότι η Απονία ε, υπογράφει ε, τις 100 συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών. Αν αυτό γίνει δεν θα υπάρχουν πλέον εμπόδια και θα ανοίξει η Απονική αγορά για την Ευρώπη. Άλλο παράδειγμα, το θέμα των πολύ αποτελεσματικών και αποδοτικών αυτοκινήτων. Εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επιβεβαίωσε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ότι θα μειωθούν στο 0,85% οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος μέχρι το 2020 ε, και επιβεβαίωσε και ποιες πρόοδοι έχουν γίνει μέχρι στιγμής και ποιες πρόκειται να προωθηθούν. Στην Ιαπωνία όλα αυτά δεν ισχύουν. Εκεί ε, υπάρχει μία προώθηση η οποία αποβλέπει μόνο την προδιαγραφή ε, ε, η Ιαπωνία 08 και βλέπουμε ότι προωθεί στα ίδια επίπεδα τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιριών οι οποίες επιτρέπεται να εισέλθουν στην ιαπωνική αγορά. Και δεν υπάρχει η δυνατότητα να, για τους Ευρωπαίους να ε, εγκαταστήσουν εμπορικές επιχειρήσεις ε, ε, στην Ιαπωνία ή εργοστάσια διότι υπεύθυνε για αυτές είναι οι περιφερειακές αρχές και βλέπουμε ότι ναι να ανοίγουμε μία αγορά αλλά τυπικά αλλά ουσιαστικά δεν επιτρέπουμε ούτε να ανοίξουμε ανοίξουν εργοστάσια ή εργαστήρια ούτε να εγκατασταθούν εμπορικές επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να πετήσουμε από την Ιαπωνία να δώσει ένα σαφές σήμα για να επιτρέψει μια πραγματική είσοδο στην ιαπωνική αγορά. Και γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε σαφείς ιδέες για το τι πρέπει να κάνουν ε, πολιτικά και οικονομικά οι εταίροι μας αλλά θέλουμε να ε, μπορέσουν στα πλαίσια αυτά να εγγυηθούν ότι θα υπάρξει άρση των μη δασμολογικών εμποδίων στις διμερείς μας σχέσεις. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σύντομα σε σχέση με τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Αντιλαμβάνομαι από όσα είπαν ε, οι συνάδελφοι με τις άλλες ομάδες που το πάνε. Όμως, αυτό το οποίο θεωρούμε ότι ισχύει είναι ότι μας συμφέρει να αρχίσουμε τις επανατεύσεις. Το νωρίτερο δυνατόν. Και νομίζω ότι κατά αυτές τις διαπραγματεύσεις, τα προβλήματα, οι επιφυλάξεις, όλα τα θέματα θα τα προχωρήσουμε. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς μπορούμε κάποια στιγμή να δούμε πώς πάνε τα πράγματα ανάλογα με το τι κάνει το το, η άλλη πλευρά, τι κάνει η Ιαπωνία. Μπορούμε πάντοτε να ε, φρενάρουμε τις εξελίξεις. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να μην ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Και επίσης, να μην ξεχνούμε ότι πρόκειται περί του αμοιβαίου συμφέροντος. Πάντοτε έχει εναλλακτικέ η Ιαπωνία. Άρα, να μην στριμωχνόμαστε μόνοι μας και έτσι να μην μπορούμε να βρούμε ε, λύσεις. Γι' αυτό σας λέω, συμφωνώ με τον εισηγητή και πιστεύω και το ένστικτό μου μου λέει, όπως και, για... Ε, όπως αυτό το τοπίο που το πρεσβεύει, όλοι μας υπό ομάδα, να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και τότε θα τα βρούμε στην πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ για τους πρασίνους. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, we welcome the opening of negotiations with... Um, και οι πράσινοι πρεσβεύουμε ότι, πρέπει να αρχίσουν να με την Ιαπωνία και έχουμε εδώ στο σχέδιο κειμένο κάποια που δεν, σημεία που δεν είναι σαφή σε σχέση με την δεσμευτικότητα. Ε, κοιτάξτε, κάθε κείμενο διεθνούς συμφωνία σύμφωνα με την ε, συνθήκη της Βιέννες για τις διεθνείς συμφωνίες, ε, ε, ορίζεται εκεί σαφώς ότι πάσα διάταξη είναι νομικά δεσμευτική. Όπως και η διαδικασία επίλυση των διαφόρων. Και επομένως τώρα προβληματίζομαι για το άλλο θέμα. Ότι ο μηχανισμός τέτοιο σε μια συμφωνία ελευθερών εμπορίου σημαίνει ότι η δικαιοδοσία ε, εκτός δημοκρατικού καθεστώτος μας οδηγεί σε κάποιες αποφάσεις, σε κάποιες ερμηνείες οι οποίες βεβαίως θα δεσμεύουν τους προσυπογράψαντες και πρόκειται για έναν ε, μηχανισμό διαιτησίας ή επιδιαιτησίας, ο οποίος όμως δεν έχει σχέση με δημοκρατική διαδικασία και συνήθως αυτό χρησιμοποιείται μεταξύ νομικών πρόσωπων, μεταξύ εταιριών. Γιατί να μην παραπέμψουμε σε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει όπως ο μηχανισμός επιλογής διαφορών του ΠΟΕ, αυτό θα ήταν ε, αρκετό. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό θα ήταν να έχουμε μια δεύτερη, δεύτερη συμφωνία, δεύτερη φάση τέλος πάντων ολοκλήρωσης της συμφωνίας όσον αφορά την, ε, την ε, μελέτη αξιολόγηση επιπτώσεων. Αν τον πάρει τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much for this to, to... Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα να απαντήσω. Εν γέννη, ευπρόσδεκτο το ψήφισμα. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικές οι διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία. Ξεχωρίζει η Ιαπωνία σε σχέση με άλλες διαπραγματεύσεις. Η Ιαπωνία θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και τις συνθήκες. Δύσκολο να απαντήσω. Πρέπει να δούμε πρώτα το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Βλέποντας τα στοιχεία τα διαθέσιμα, και την αξιολόγηση αντιχτύπου συνεπιών που θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα. Βλέπουμε ότι μια φιλόδοξη φωνή από την Ιαπωνία μπορεί να είναι υποφελής στο ύψος του 1% του ΕΠ. Είναι ένα από τα καλύτερα μέσα που έχουμε στο χέρι μας για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Συμφωνώ ότι δεν θα είναι εύκολε οι διαπραγματεύσεις. Πρέπει να μπούμε έτοιμοι, ετοιμασμένοι, για να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους. Ευπρόσδεκτα τα σχόλια που ακούστηκαν. Θα αναφερθώ σε μερικά από αυτά. το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής γίνεται παραλληλισμός μεταξύ εξάλληψης δασμών και εξάλληψης μη δασμολογικών φραγμών. Η Ευρώπη δεν θα μειώσει με άλλα λόγια τις, τα μέτρα προστασίας της αν δεν κάνει το αντίστοιχο η Ιαπωνία. Παράλληλα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις. Δεν θα μειωθεί η προστασία συγκεκριμένων τομέων στην Ευρώπη αν δεν γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ιαπωνία. Είμαστε έτοιμοι να αναστείλουμε τις διαπραγματεύσεις αν η Ιαπωνία δεν κάνει αυτά που υπόσχεται. Και έχουμε θέσει χρονοδιάγραμμα. Ένα χρόνο μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Θα παρακολουθούμε από πολύ κοντά τις εξελίξεις σε συντονισμό με όλα τα θεσμικά όργανα. Αν θα συμμορφωθεί με τι υποχρεώσει τη Ιαπωνία. Εάν δεν σεβαστεί τι υποχρεώσει η Ιαπωνία, θα κάνει τα δέοντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πάμε μάτια τα χέρια στις διαπραγματεύσεις. Πάμε με επιθετικά μέσα, αλλά και αμυντικά. Έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα αντιστοιχεί στις φιλοδοξίες μας. Θα είναι κάτι επωφελές για, τον, για τους ευρωπαϊκούς λαούς. για σαφές χρονοδιάγραμμα για την εξάλληψη δασμών, δασμολογικών φραγμών, αυτό είναι κομμάτι των διαπραγματεύσεων είναι πολύ δύσκολο να το ξεκαθαρίσουμε πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό το εγχείρημα βολιδοσκοπήσεως ε, ήταν και το πλέον φιλόδοξο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δημιούργησε μια βάση. Πάνω σε αυτή μπορούμε να οικοδομήσουμε κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων για να πετύχουμε σαφές χρονοδιάγραμμα. Και όπως προανέφερα, αυτό κινείται παράλληλα με εξάλληψη δασμών. Θα εξετάσουμε το θέμα φορολογικών και, ε, κινήτρων, καινοτόμο αυτό για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου για τα αυτοκίνητα και συγκεκριμένη δέσμευση της Ιαπωνίας που αναλύθηκε στις πρώτες επαφές. και δέσμευση για διευκόλυνση το συστήματος διανομή σε διάφορες περιοχές και διανομή αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία της Ιαπωνίας. Υπάρχουν ανησυχίες και από πλευράς Ιαπωνίας και πλευράς Ευρώπης. να μην παρισφρήσουμε στις ε, συνταγματικές εξουσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας. Αυτό ισχύει και την Ευρώπη και την Ιαπωνία. για την διευθέτηση των διαφορών. Και αν πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο στον ΠΟΕ. Αυτό θα είναι περιπλοκότατο, αν όχι ανέφικτο, διότι αυτές είναι άλλου είδους συμφωνίες. Το να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στη διευθέτηση των διαφορών θα προβλέπεται από τη συμφωνία είναι σίγουρα με της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα το σκεφτούμε όντως. Δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις για όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είμαι ακόμα επίτροπος δυστυχώς. Για την Ταϊβάν, άριστες οι διμερείς μας σχέσεις με την Κινέζικη Ταϊπέ Έχουμε ομάδες εργασιών που δίνουν αποτελέσματα. Υπάρχει μία που ασχολείται με τη διευκόλυνση ε, και πρόθεση του διμερούς εμπορίου. Ευχαριστώ για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Ο εισηγητής ο Μάρτιν Κάζακ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ τους συντονιστές, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά που ανέφερε, τις προσδοκίες που υπάρχουν, την αξιολόγηση που έκανε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία. Μοιράζομαι και εγώ τις ανησυχίες και αυτά που υπόθηκαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά είμαι πεπισμένος ότι μια τέτοια συμφωνία είναι προς όφελος θα είναι πολύ υποφελής τώρα αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν παγκόσμιος φορέας οικονομικός και πολιτικός, μεγάλης εμβελίας, θα πρέπει να διαπραγματεύεται ε, με μια τόσο μεγάλη δύναμη όπως η Ιαπωνία. Παρά όλες τις δυσκολίες που ίσως αντιμετωπιστούν, Πρέπει να γίνει κάτι. Όταν είναι εκεί και πηγαίνει μια ευρωπαϊκή εταιρεία και πάει στην Ιαπωνία, έχει προβλήματα. Το είδαμε τα μάτια μας, τα πήγαμε εκεί σαν ε, αντιπροσωπεία όμως ότι υπάρχουν πολλές πετυχημένες ευρωπαϊκές εταιρείες που τα καταφέρουν μια χαρά στην Ιαπωνία. Και βγάζουν κέρδη στην Ιαπωνία. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, σαφές χρονοδιάγραμμα για να ξεπεραστούν οι δεσμολογικοί και μη δεσμολογικοί φραγμοί πιστεύουμε ότι είναι κάτι απαραίτητο, χρειάζεται χρονοδιάγραμμα, σαφές, με δεσμεύσει από τις δύο πλευρές και κυρίως την Ιαπωνία. Γι' αυτό στο ψήφισμα επιμένουμε για μία ρήτρα συγκεκριμένη για αναθεώρηση. Με αυτή τη ρήτρα περιοδικά μπορούμε να αναθεωρούμε το βαθμό στον οποίο πληρούνται αυτές ε, οι προδιαγραφές, κατά πόσο μορφώνται με τι υποχρεώσει του. Θα πρέπει να υπάρχουν οδικοί χάρτες, προσανατολισμοί για να γίνουν σεβαστέ αυτές οι δεσμεύσει. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ευαισθησίες για διάφορους τομείς, όπως είναι η βιομηχανία. Εγώ, με τον κύριο Λάγκε, με τον κύριο Κασπάρη, μπορούμε να συζητήσουμε μήπως υπάρξει και άλλη παράγραφος που θα εστιάζεται επί συγκεκριμένης πτυχής, κυρίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ούτω ώστε να έχουμε τα απαραίτητα χέγγια ότι οι αναληφθήσεις υποχρεώσεις θα τηρούνται. Πριν από δύο μέρες, η ομάδα του ΕΛΚ διοργάνωσε ειδικό σεμινάριο με τις επιχειρήσεις με θέμα αυτή τη συμφωνία και από ό,τι γνωρίζω όλοι οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ήταν υπέρ της συμφωνίας εκτός από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Όμως θεωρώ ότι τώρα είναι η στιγμή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει αυτή τη δυνατότητα, να δημιουργήσει τη δυνατότητα για μια πλήρη συμφωνία που είναι υποφελής για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. θα δημιουργήσει πολλές δυνατότητες, πολλές ευκαιρίες με τέτοια συμφωνία. Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για όλους. Σα ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ για τη ζωή συζήτηση, λέει ο Προέδρο. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών η 18 η Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Να ρωτήσω κάτι. Δεν μπορώ να μείνω μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Οπότε, οπότε θα αντικατασταθώ στην Προεδρία. Έχω όμως ακόμη ε, δύο θέματα επί των οποίων είμαι εισηγητής και θα ήθελα να μπορέσω να τα παρουσιάσω για να μπορέσω συνέχεια να εγκαταλείψω τη συνεδρίαση. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, σας ευχαριστώ. Προχωρούμε λοιπόν τώρα στο 34 και 35 που είναι συνδεδεμένα διότι το ένα αναφορά την συμφωνία μεταξύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη και την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με αυτή τη συμφωνία διότι τον Ιούνιο υπογράψαμε τη συμφωνία με τη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη ε, σχετικά με τις παραχωρήσεις όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών βάσει τη συμφωνία του ΓΚΑΤ ε, για να αντιμετωπιστούν οι ε, αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ε, ε, ε, βιομηχανία πουλερικών και είδαμε ότι υπάρχουν ε, ε, εξαγωγείς οι οποίοι εποφελούνται από το κενό και ε, παρήγαγαν κρέας το οποίο δεν σεβόταν το μίνιμουμ 54% και γι' αυτό επειδή η Βραζιλία και η Ταϊλάνδη ήταν οι χώρες οι οποίες είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της αγοράς υπήρξε μια αναδιαπραγμάτευση ε, της συμφωνίας κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. Δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να το δεχτούμε. Ε, να δεχτούμε δηλαδή να, να υπάρξει αυτή η τροποποίηση διότι έτσι θα επιληθούν τα, οι δυσκολίες ε, οι οποίες ε, μπορεί να αντιμετωπιστούν. Είναι δηλαδή μία συγκροτημένη προσέγγιση. Καταρχήν πρέπει να προστασία της δικιάς μας ε, ε, βιομηχανίας για να αποφύγουμε την παράκαμψη των, ε, της επιβολής δασμών. Και από την άλλη πλευρά η, οι εταίροι μας θα πρέπει να καλύπτονται και αυτοί σχετικά με τις ποσοστώσεις και τους δασμούς. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα σύνολο στη συμφωνία με παραχωρήσεις οι οποίες να καλύπτουν και τις δύο πλευρές ε, αυτές είναι οι απόψεις μου θα παρουσιάσω ένα σχέδιο εκθέσεως αλλά αυτά είχα να σας πω σαν πρώτα σχόλια και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσω ε, να το προχωρήσω. Ο ε, κύριος Στράσερα από το ΕΛΚ. Νομίζω ότι πολύ σωστά κύριε Πρόεδρε λέει ο κύριος Στράσερ τονίσατε ότι το 34 και το 35 ε, θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι παρεμφερή το 34 συγκεκριμένα αναφέρεται στην ε, πρόληψη των ε, παραβιάσεων των ε, εισαγωγέων κρέατος προς την Ευρώπη και στο σημείο 35 ασχολούμαστε με την ε, βελτίωση του κανονισμού σχετικά με την δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Εγώ εκ μέρους μου μπορώ να συμφωνήσω με τα συμπεράσματά σας και θα σας στηρίξω. Ευχαριστώ. Ε, πάλι ο κύριος Κλάρκ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, συμφωνούμε πλήρως με τις παρατηρήσεις σας και τα συμπεράσματά σας, διότι όπως είπαν και οι συνάδελφοι έχουμε εδώ δύο θέματα, τις συμφωνίες και διαπραγματεύσεις για το κρέας πουλερικών με τη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη και ε, ε, την ε, συμφωνία σχετικά με το επίποδο των τελωνιακών δασμών. Ο ΠΟΕ μπορεί να υπάρξει, μπορεί να δεχθεί μία αύξηση των δασμών εάν υπάρξει έξαρση των εισαγωγών, αλλά ζητά από τις ε, ε, χώρες που εξάγουν τα προϊόντα να επανισορροπήσουν τις ε, υποχωρήσεις που τους έχουν γίνει και αυτό γίνεται εδώ με τη Βραζιλία και την Ιλάνδη όπου θα να διαπροσδιοριστεί ο τελωνιακός θεσμός ε, και ε, σύμφωνα με τις αρχές του ε, ΠΟΕ θα υπάρξουν και αντισταθμιστικές υποχωρήσεις. Είναι ένα σύνηθες αίμα από πλευράς διαδικασίας του ΠΟΕ αλλά χρειάζεται την αποδοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι θα μας την χορηγήσετε. Ευχαριστώ ευχαριστώ. Η η υποβολή του, της συστάσεως θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση 17 και 18 του Σεπτεμβρίου. Ε, έτσι ολοκληρώσαμε την εξέταση των θεμάτων μας. Σας εύχομαι καλές διακοπές και ελπίζω να περάσατε καλά όπως πέρασα και εγώ. Στη συνέχεια θα με αντικαταστήσει ο Αντιπρόεδρος και ε, ε, θα εξετάσετε τα υπόλοιπα θέματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ε, ε, τώρα θα συνεχίσω τη συνεδρίαση και ερχόμαστε στο σημείο 32. Σχετικά με την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο θέμα των εμπορικών συναλλαγών και επενδύσεων και δίνω το λόγο στον εισηγητή κύριο Σαραντήλ. Για να σας τα πω στην μητρική μου γλώσσα. Παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά Tak, vážení kolegové, vážené kolegyně, ten té navrhované zprávy už sám o sobě. Κυρίες και κύριοι, η έκθεση αυτή αφορά στην πρόσβαση που πρέπει να έχουν οι ΜΜΕ σε δάνειο, σε πίστοση, κυρίως όταν επιχειρούν εκτός ΕΕ. Να μην αρχίσουμε τώρα τα ενιολογικά, τα συμμεσολογικά σε σχέση με τον ορισμό της ΜΜΕ, γιατί αυτά τα έχουμε συζητήσει, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Κατά τη γνώμη μου, εδώ, στο πλαίσιο αναφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ΜΜΕ σημαίνει μια εταιρεία που δεν ανήκει σε κάποιο όμιλο εταιρεών, υπερεθνικό, πολυεθνικό, έχει πάνω από 15 ε, εργαζομένους και κύκλο εργασιών έχει μέχρι 50, ε, 50 εκατομμύρια ετησίως. Ε, τώρα, αυτό είναι κάπως αφαίρετο. Έχουμε άλλωστε και τις μικροεπιχειρήσεις. Οι μικροεπιχειρήσεις είναι οι πραγματικά μικρές επιχειρήσεις που έχουν κάποιους εργαζομένους, ας πούμε, 12, περίπου Τέλος πάντων, για τους σκοπούς της εκθέσεώς μου αυτός ο ορισμός αρκεί. Τώρα, στην εσωτερική αγορά έχουμε 23 εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσεις που λειτουργούν. Απασχολούν σχεδόν το 75% των εργαζομένων στον δυτικό τομέα. Και δημιουργούν το 80% των δημιουργουμένων θέσεων απασχόληση. Όμως, μόλις 25% αυτών των ΜΜΕ επιχειρούν εκτός συνόρων. το συνόρων της χώρας εγκατάστασης. Και μόνο 13% εκτελούν συναλλαγές εκτός τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός της ενιαίας αγοράς. Δηλαδή σε μια άλλη αγορά κάπου στον κόσμο. Προσπαθούμε εδώ τώρα να διερευνήσουμε τους λόγους αυτού του φαινομένου. Να δούμε πώς οι επιδόσεις μας μπορούν να βελτιωθούν. Η λογική τι λέει. Ότι εάν σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε διεθνή κλίμακα δραστηριοποιηθούν οι ΜΜΕ, αυτό θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Οπότε, θεωρούμε ότι πρώτα πρώτα η έλλειψη ενημέρωσης και πληροφοριών και δεύτερον η έλλειψη χρημάτων οδηγεί σε αυτή την απουσία των ΜΜΕ από τη διεθνή σκηνή. Θα πρέπει επομένω να δούμε τι γίνεται με κάποιο είδους ε, νέε δομέ διοικητικέ, γραφειοκρατικές που να υποστηρίξουν τι επιχειρήσεις μας. Τι ισχύει σήμερα. Αυτό το οποίο ισχύει σήμερα ο μηχανισμός που υπάρχει σήμερα είναι ανεπαρκής. Άρα, οι πληροφορίες να είναι κάπως συγκεντρωμένες για το τι ισχύει στην παγκοσμία αγορά και έτσι να μπορούν να βρουν το δρόμο τους, να μπορούν να προστατολιστούν, να μπορούν να κινηθούν στη διεθνή αγορά οι επιχειρήσεις μας. Επίσης, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να έχουν περισσότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Έχουμε κάποια προγράμματα βέβαια τα οποία είναι μέρη καλύπτουν τα προβλήματα αυτά. Έχουμε ένα σωρό χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε ένα πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα, έχουμε διάφορα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και όλα αυτά που σκοπούν στο να ε, τις, βοηθήσουν. Έχουμε βέβαια και κάποιους πόρους που έρχονται κατευθείαν από τον κοινωνικό προπολογισμό, όμως τίποτα από όλα αυτά δεν ασχολείται, δεν αποσκοπεί στην άμεση υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διεθνή σκηνή ούτε βοηθά σε επενδύσει στον ίδιο χώρο. Επομένω, θα πρέπει να δούμε τώρα τι είδου εμπορική πολιτική, τι είδου επενδυτική πολιτική ε, μπορούμε να κάνουμε, διότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Άρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να έχουμε τέτοιου είδου άσκηση πολιτική. Τέτοιου είδου πολιτική να φτιάξουμε και επομένω θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβληματιστεί, να σχεδιάσει ε, κάποιο είδους ε, ε, μέσο εργαλείο για να βοηθήσει τις εξαγωγές. Το ονομάζω Export Facility στα αγγλικά, στο EU Exim, το λέω στο κείμενό μου. Και αυτό επομένως να δραστηριοποιείται σε κάθε χώρα μέλος, να βοηθά στις, στις εξαγωγές, και τέλος πάντων να υποστηρίζει τις ήδη λειτουργούσες ε, ΜΜΕ. Επίσης, έχω εδώ πέρα ένα κατάλογο από τις ε, ενδεχόμενες, τις δυνατές ε, επιχειρήσεις, τις δυνατές υπηρεσίες, που αυτό το εξήμ, αυτό το, αυτή η διευκόλυνση θα μπορούσε να καλύψει και να προσφέρει. Βεβαίως και θα μπορούσε κανείς να να, να, να, να κόψει κάποιε αυτέ τι υπηρεσίε ή και να προσθέσει άλλε, ανάλογα με το τι θέλουν οι συνάδελφοι, τι θέλουν πολιτικέ ομάδε. Δεν θέλω τώρα να κάτσω να, να σα πω λέξη προ λέξη τι λέει το κείμενό μου. Αυτό με όλο το σεβασμό που το κάνετε κι εσεί. Όμω, θέλω να σα τονίσω για άλλη μια φορά ότι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε την οικονομία της Ευρώπης στη συγκυρία αυτή της κρίσης. Διότι θεωρώ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα πρέπει, όπως είπα στην αρχή, να καταλάβουμε ότι οι δραστηριότητες αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκτός Ευρώπης είναι περιορισμένοι. Άρα, θα πρέπει να άρουμε αυτούς τους περιορισμούς, θα πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ. Αυτά από πλευράς εισήγησή μου και περιμένω πώς και πώς τις παρατηρήσεις σας, συνάδελφοι. Και βεβαίως όποιος έχει κάτι επικοδομητικό να εισφέρει, να αλλάξει στο κείμενο και αυτό επίσης είναι καλοδεχούμενο. Ελπίζω ότι να τα βρούμε, να καταλήξουμε σε κάτι που θα συγκεντρώνει τη Γενική Συνένεση. Ε, ελπίζω να επιψηφιστεί και εδώ και στην Ολομέλη έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και τώρα δίδω τον λόγο καταρχήν στους κοιόδης εισηγητές και καταρχήν στον κύριο Κουαρέρα Σαμόρα. Συγκυρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ως εισηγήτρια, σκιώδης, θα ήθελα να σας πω τις παρατηρήσεις μου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, θα πρέπει να ωφεληθούμε από την προτέρα εμπειρία των κρατών μελών για τι ΜΜΕ. Επίση θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ό,τι και να γίνει ε, σε σχέση με την υποστήριξη των ΜΜΕ θα πρέπει αυτό να αποτελεί μια προσθέμενη αξία, πρέπει να είναι συμπληρωματικό των όσων ήδη ε, ισχύουν. Θα πρέπει επομένω να, να, να παραμείνουν, θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν τα προγράμματα τα οποία ήδη ισχύουν. Οπότε, στα, πλαίσια αυτή τη υποστήριξη των ΜΜΕ θα πρέπει να δούμε πώς θα δεσμευτούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ίδιες χείουσες πολιτικές των κρατών μελών και αυτό να γίνει σε όλα τα επίπεδα. προσθέμενη αξία θα είναι μια πολιτική ευρωπαϊκή που να έχει την υποπτία, να έχει την αξιολόγηση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε τις καλύτερες των πρακτικών που υπάρχουν και με αυτόν τον τρόπο όντως να μην αξία και θα πρέπει να δούμε ότι η χρηματοπιστωτική κρίση υπέσκαψε τα χρηματοδοτικά μέσα για την πρόσβαση σε, σε, σε, σε που χρειάζονται για τη λειτουργία τη Οπότε, για να μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάτι να κάνουμε, να έχουμε παραπάνω πόρους, να έχουμε καλύτερα συστήματα, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ ε, στην διέξοδο από την κρίση. Όμω αυτό ακριβώ να αποσκοπεί στο να διεθνοποιηθεί η δραστηριότητα των ε, επιχειρήσεων αυτών. Αυτό αναμφίβολα και των ΜΜΕ και κάθε επιχείρηση θα βοηθήσει στο να έχουμε ανάπτυξη οικονομική και απασχόληση. Ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες διεθνώς και κυρίως στις αναδυόμενες οικονομίες. Και να δούμε πώς θα επιλύσουμε αυτές τις δυσκολίες που οι ΜΜΕ και οι μικροεπιχειρήσεις ε, στις οποίες προσκρούν. Οπότε να δούμε τι θα γίνει πέραν το, το, της ενιαίας αγοράς που φυσικά είναι πάντα την προτεραιότητα. Είναι κατακλείδη. Θέλω να πω στον εισηγητή ότι είμαι διατεθειμένη να τον βοηθήσω όσο γίνεται στο έργο του. Ευχαριστώ. Η, η συγγήτρια των σοσιαλιστών δεν παρίσταται, οπότε επιτρέψτε μου να κάνω μία παρατήρηση. Νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να εστιαστούμε στα μηνύματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιζητήσουμε σε άλλες χώρες εταίρους με τους οποίους να μπορούμε να διοργανώσουμε ε, εκδηλώσεις ε, για επαφές και ε, να, επισημαίνουμε ε, την γραφειοκρατία των άλλων κρατών δηλαδή να υπάρχει μία ε, σωστότερη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για λογαριασμό των μικρομεσών επιχειρήσεων και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Μάρφη που έχει σχόλια. Uh, λοιπόν, κανονικά περνάει από του συντονιστέ των πολιτικών ομάδων ε, η διαδοχή των ομιλιών διότι αυτό γίνεται με τις πολιτικές ομάδες όταν είναι ο κύριος Ντογκιούχτε εδώ αλλά είσαστε εσκι... εσείς δεν μου φανήκατε ε, ότι είστε ε, σκιώδης εισηγητής γι' αυτό και ζήτησα πρώτα να παρέμβουν οι σκιώδης εισηγητές και μετά οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές άρα ε, έχω σημειώσει την αίτησή σας να παρέμβετε δεν ήταν αυτό όμως που εγώ ότι ε, ε, δεν ήταν ο στόχος τη παρεμβάσεώς μου, νόμιζα ότι είχατε ε, τελειώσει με τους σκιώδη ε, και γι' αυτό ζήτησα το λόγο. Αλλά είναι ένα νέος κόσμος. Όχι, πρώτα δίνουμε το λόγο στους εισηγητέ. μετά στους σκιώδη εισηγητέ. Από τη δικιά σας πολιτική ομάδα κανείς δεν με ενημέρωσε ότι είσαστε σκιώδη εισηγητή. Αν είστε ε, οι εισηγητές, πέστε μου τον και θα σας δώσω τον λόγο στη σειρά των πολιτικών ομάδων που θα παρέμβουν. Τώρα όμως έχω μόνο δύο σκιώδεις εισηγητές, την κυρία Κορέρα Σαλμόρα, την κυρία Μπαλζάνη. Άρα αυτές θα παρέμβουν πρώτες και μετά θα δώσω το λόγο σε όλους τους υπολείπους. Οπότε με τα βεβαιότητα, θα μπορέσετε να παρέμβετε όταν το επιθυμήσετε. Τώρα όμως οι πρώτοι που ζήτησαν το, ο πρώτος που ζήτησε το λόγο και όχι ο σκιώδης εισηγητής είναι ο κύριος Μέρφυ ο οποίος θα καταγραφεί στη λίστα των περαιτέρων ομιλητών. Ωραία. Προ, προσβλέπω στο χώρο που θα μιλήσω. <laughs> Η κατάσταση είναι σε πολλές χώρες όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις στην Ιρλανδία. Τον τελευταίο χρόνο πέντε εταιρείε έκλειναν κάθε μέρα κατά μέσο όρο. Περισσότερες από αυτές είναι μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό συμβαίνει όχι διότι δεν υπάρχει επαρκής διεθνής παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν έχουν πρόσβαση σε πιστώσει κυρίως για να έχουν διεθνή παρουσία αλλά σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στην κατάρρευση τη καταναλώση των καταναλωτών σε πολλέ χώρε. Έχει μειωθεί στην Ιρλανδία 15%. Είναι άμεσα αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητα που επιβάλλονται και η λύση στην κρίση σύμφωνα με του ηγέτε μα είναι περισσότερη λιτότητα και αυτό θα χειροτερεύσει την κατάσταση στους εργαζομένους, άρα για τους καταναλωτές, άρα μεγαλύτερη κρίση για τις μικρές επιχειρήσεις. Δευτερεύον παράγων, σημαντικός, πολύ σημαντικός, είναι η έλλειψη πρόσβαση στην πίστοση. Συμφωνώ με αυτό. Όχι μόνο για διεθνή παρουσία, αλλά για οτιδήποτε άλλο. Πολλέ μικρέ επιχειρήσει δεν έχουν πρόσβαση σε πιστώσει για να κάνουν οτιδήποτε πλέον. Και υποφέρουν. Έχουν, ε, τους πνίγει αυτό. Και αυτό είναι, οφείλεται στο ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα. Αντιλούνται δεκάδε δισεκατομμύρια δημοσίου χρήματο, ευρώ, 3 ε, ευρώ να περνάνε από το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα και δεν πηγαίνουν σε δανεισμό μικρών επιχειρήσεων για την άψη της ε, οικονομίας κλπ. Απλώς θέλουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος οι τράπεζες πηγαίνοντας αγοράζοντα ομόλογα των χωρών που δέχονται επιθέσεις των αγορών ή απλώς ξαναμπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα αυτή φίλεται στο ιδιωτικό είναι κλειοδότημα του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματο, άρα χρειάζεται να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι συνδυασμό ιδιωτικού δημόσιου τομέα, τραπεζικό σύστημα, για να δίνει πιστώσει στι μικρέ επιχειρήσει. Η λύση στην κρίση, πιστεύω, δεν είναι η διεθνοποίηση σε μια παγκόσμια οικονομία που αντιμετωπίζει και αυτή η κρίση. Θα μπορούσε να έχει μικρό αποτέλεσμα, αλλά η λύση θα πρέπει να σταματήσει τα μέτρα λιτότητα και θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατικό έλεγχο τραπεζικού συστήματο. Όσον αφορά για το μέσο για εξαγωγές, εισαγωγές, κατά χώρα, από πού θα προέλθουν οι πόροι, πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, συγκεκριμένη πρόταση. Αν δημιουργηθεί ένα τέτοιο μέσο, ένα τέτοιο εργαλείο, για να υπάρξει πρόσβαση σε αυτό το μέσο, ο όρος θα είναι να μην υπάρχει προς τα έξω ανάθεση της παραγωγής. Αυτά που παράγονται στην Ευρώπη να μην μεταφερθούν εκτός Ευρώπης σε παραγωγή μετά για να δημιουργηθεί πίεση προς τα κάτω των αμοιβών, πραγματικά θα πρέπει να είναι μια επέκταση στους αγορές και αύξηση της παραγωγής πραγματική. Θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για πρόσβαση στο μέσο αυτό. Ευχαριστώ. Um, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνήσαμε στην πολιτική μου ομάδα χτες το βράδυ ότι θα είμαι σκιώδης για την έκθεση, για την ομάδα μου Όλοι το ξέρουν τώρα. Ζητούμε συγγνώμη που το ρυθμίσαμε νωρίτερα. Γενικά τώρα. Οι πράσινοι πιστεύουν ότι χρειάζεται προσοχή όσον αφορά τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διεθνοποίηση είναι πολύ δαπανηρή, δύσκολο να τη χειριστεί κανεί. Χρειάζεται ανθρώπινου πόρου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα για να αναπτυχθούν καλύτερα αγαθά σε τοπικό επίπεδο και υπηρεσίες. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις επενδύουν πολλά χρήματα για να έχουν διεθνή παρουσία στις επιχειρήσεις τους, αλλά αποδυναμώνονται στην προσπάθεια αυτή και αποτυχάνουν. Για τους σκοπούς της έκθεσης, στην γνωμοδότηση Winkler για την ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέρονται δύο σημεία που θα θέλαμε να ληφθούν υπόψη τον εισηγητή στο σχέδιο έκθεση. Ποια είναι αυτά. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν διεθνοποίηση να προστατεύονται από αθέμητες εμπορικές πρακτικές από χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέσα για προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στις αγορές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί για να έχουν ευκολότερη πρόσβαση ε, στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές των εμπορικών εταίρων. Ευχαριστώ. Και τώρα ο επόμενος ομιλητής. Τώρα έχετε το λόγο. κύριος Μος. Πρώτα πρώτα. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον εισηγητή. Είναι σημαντικό το ότι ασχολήθηκε με αυτό τον κλάδο της οικονομίας. Και Μα επέσε την προσοχή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο παράγραφο ότι δηλαδή 75% των θέσεων εργασία στον ιδρυτικό τομέα πρόκειται από ΜΜΕ και αυτό έχει βοηθήσει. Ε, δηλαδή ο κλάδο αυτό βοήθησε στη δημιουργία του 80% των νέων θέσεων εργασία και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτέ οι ΜΜΕ να μπορέσουν να καταλάβουμε, να μπορέσουμε εμεί να καταλάβουμε ότι δεν ακολουθούν την οικονομία. Είναι ατμομηχανίτε και προέκυψε τα τελευταία χρόνια ότι η αριστερά με την εξαίρεση του κυρίου Μέρφη η παλιά αριστερά, η κλασική αριστερά, η παραδοσιακή αριστερά επιτίθεται στις επιχειρήσεις, τις μεγάλες κυρίως και τι είδα σήμερα το πρωί ότι η Πεζό έχει 200 εκατομμύρια σημείες μηνιαίως. Και μιλάμε για 6.500 θέσει που θα χαθούν και στην ε, Γαλλία. Υπάρχει τεράστια πίεση να υπάρξει κάποιο σχέδιο διάσωσης της πεζό. Και αυτά τα χρήματα της διάσωσης φυσικά θα επέθαν στην οικονομία, θα δημιουργούσαν θέσεις εργασία. Ανέκαθεν επομένως η κέντρο δεξιά ήταν κατά των εθνικοποίησεων και κυρίως των κρατικοποίησεων και εθνικοποίησεων των τραπεζών. Έχει δίκιο ο κύριος Α, σήμερα κατ' εξαίρεση συμφωνώ, είδατε σε πόσα πράγματα μαζί του. Ότι η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε στο να μην υπάρχουν πια δάνεια, πιστώσεις και, και φυσικά αυτό ισχύει και για τα δάνεια προς τις ε, ΜΜΕ. Οπότε, επομένως, είναι βάσιμο το να έχουμε κάποιο είδους ε, κυβερνητική ενέργεια ε, προς αυτό το σκοπό, πώς να τους χορηγηθούν δηλαδή κάποιες πιστώσεις των ΜΜΕ. Τώρα, η έκθεση μας οδηγεί στο ότι αξίζει κανείς να ασχοληθεί με τον προβληματισμό αυτό. Το ότι δηλαδή καλύτερα αυτά όλα να γίνουν από την Κομισιόν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση παρά σε επίπεδο κρατικό. Το λέει και εδώ πέρα κάπου η έκθεση που λέει ότι για αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν για την ανταγωνιστικότητα. Το κέντρο τη είναι είναι κάπως αδόκη μετάφραση και λέει εδώ πέρα ότι έχουμε ένα κορβανά 2,5 δι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα δει αυτά για να μας τα επιβεβαιώσει η Κομισιόν. Αυτό τι είναι. Υπάρχει αυτός κορβανάς ή μήπως, τι είναι, είναι ευσεβής πόθος, είναι κάποιο σχέδιο προς Πέραν αυτόν πάντως. Αυτή καθ' αυτή η ιδέα, το ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλία θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο κομισιών, κάτι γνώμη μου στερείται νοήματος. Είναι χαμένος χρόνος. Ο συγκριτής είναι Τσέχος. Η οικονομία της χώρας του είναι πολύ πετυχημένη, πολύ υγιής. Έχετε τέτοιες επιχειρήσεις στην Τσεχία, που μπορεί να έρθει εδώ στις Βρυξέλλες να τραβήξει την προσοχή κάποιων υπαλλήλων της Κομισιόν όταν δεν είναι σε διακοπές. Δεν νομίζω. Ε, όσο κάνουν ε, σε ένα χρόνο διακοπές πάλι της Κομισιόν, εγώ τα κάνουν σε δέκα χρόνια. Τέλος πάντων, νομίζω ότι καλύτερα να γίνουν όλα αυτά που λέει έκθεση σε εθνικό επίπεδο. και οι επενδύσει και το εμπόριο είναι αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω λέει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Και εμεί όμω πάγια λέμε ότι η συνθήκη αυτή δεν έχει δημοκρατική νομιμότητα. Κυρίω όσον αφορά τη χώρα μου και οι ΛΥΠΔΕΜ, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, Δημοκράτες, ακούστε να δείτε, ε, υποσχέθηκαν δημοψήφισμα και μετά τα γυρίσανε. Οπότε όλα αυτά που λέτε εδώ πέρα δεν ξέρω τι να πω. Πρόεδρε, επίσης κάτι άλλο. Από τότε που άρχισε να ισχύει αυτό το σύστημα του να δίνουμε το λόγο στους ε, αγορητές, μετά τους ε, σκιώδεις ηγητές, να έχουμε προτεραιότητες σκιώδεις ηγητές, τότε εγώ για να λαμβάνω το λόγο θα είμαι κάθε φορά σκιώδης ηγητής για, για τα πάντα. Όχι, όχι, εντάξει, αυτό να το κάνετε, είναι αλλά δεν είναι καινούριο. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά ακόμη για την έκθεση αυτή και θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σύντομη, διότι εχθές Ε, μάλλον ε, έχουμε τους εκπροσώπους ε, του, της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας εδώ και καλό θα ήταν να μπορέσουμε εφόσον έχουν έρθει από το εξωτερικό να τους διαθέσουμε κάποιο χρόνο. Γι' αυτό και τώρα δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ που είναι δυνατότητα να εκφράσει απόψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα. Πολύ σημαντικό, περιπλοκότατο, συμφωνούμε με την ανάλυση που ακούστηκε για τα συμπληρωματικά ωφέλη αυξημένη διεθνού παρουσία των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν σημαίνει μόνο ανάπτυξη παραπάνω και δραστηριότητα, αλλά καινοτομία, δημιουργία δυναμικού, αύξηση παραγωγικότητας. Συμφωνούμε και με τι ανησυχίε που ακούστηκαν. Πράγματι, σε αυτή τη φάση έχουμε αυξανόμενο οικονομικό έλλειμμα, κενό. Γίνονται τα πράγματα σε πολλά κράτη-μέλη πολύ δύσκολα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύ δύσκολο να χρηματοδοτήσουν εξαγωγικές δραστηριότητες. Υπάρχουν εθνικά προγράμματα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, διάφορα μέσα για εξαγωγικές πιστώσεις. Γνωρίζουμε όμως ότι οι εμπορικές τράπεζες αποσύρονται από αυτή την αγορά σιγά σιγά, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Τι μπορεί να γίνει για τις υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλές, ενημέρωση. Χαρτογραφούμε την κατάσταση. Ξεκινάμε, είμαστε στη φάση ανάθεσης του εγχειρήματος. Έτσι, στο τέλος, τέλος του πρώτου εξαμήνου του χρόνου, θα έχουμε πλήρη ανάλυση της εικόνας στα διάφορα κράτη-μέλη, στις εξωτερικές αγορές, πώς μας συνδυαστούν οι διάφοροι παράγοντες, τι συμπράξεις μπορούν να υπάρξουν, που υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις, που υπάρχουν κενά. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τις πιστώσεις. και τα υφιστάμενα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα προτινόμενα για το επόμενο πολιτές πλαίσιο επιτρέπουν χρηματοδότηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων των μικρομεσών επιχειρήσεων. Είναι κάτι που καλύπτεται. Δεν έχουμε ειδικό μέσο για κάτι τέτοιο. Καλύπτεται όμως ως έχει οι μεσάζοντες οι χρηματοπιστωτικοί μπορούν να αναπτύξουν χαρτοφυλάκια ε, για εγγύσεις για εξαγωγικές δραστηριότητες Φερρυπίν όπως υπάρχουν προσεγγίσεις για προϊόντα που είναι οικολογικός καινοτόμα για τη μεταφορά επιχειρήσεων αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τον εισηγητή να διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής των διάφορων εναλλακτικών που προτείνονται. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο σαν ευκαιρία. Και περιμένουμε την έκθεση. Για τα 2,5 δις έχω ερώτημα. Είναι πρώτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του νέου πολιτούς πλαισίου το κόσμο που είναι για ένα πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων. 58% του ποσού αφορά τα διάφορα χρηματοσυντικά μέσα, χρήματα που, που έμεσα πηγαίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 17% είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων. 75% του κονδυλίου αφορά υπηρεσίες και χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο δίνω τώρα στον εισηγητή για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για ε, τις πολύ πολύτιμες ε, παρατηρήσεις σας και την επισήμαση για το ενδεχόμενο ε, δυνητικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Ντάρτμουθ, κύριε Ντάρτμουθ, ούτε να μ' αρέσει το, η συνθήκη της Λισαβόνας, δεν την υπερψήφισα στο Κοινοβούλιο, αλλά ισχύει, τη σέβομαι, και ε, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι αποκλειστικά αρμόδια στον τομέα του εμπορίου. Άρα δεν κάνουμε κάτι αφύσικο, δεν πάμε αντίθετα στις εθνικές αρμοδιότητες των κρατών. Είναι απλώς κάτι το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί για να μπορέσει να υπάρξει ε, μία καλύτερη αντιμετώπιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να υποχρώσουμε μία μικρομεσαία επιχείρηση να κινηθεί διεθνώς, αλλά ε, αν έχουμε ορισμένες δυνατότητες που μπορεί να τη βοηθήσουν, εάν κάποιος θέλει να τις χρησιμοποιήσει μπορεί να υποφεληθεί. Εξού και πιστεύω ότι μετά από αυτή την πρώτη εισαγωγή είμαστε σε καλό σημείο για να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα και προσβλέπω στην μελλοντική συζήτηση και σε στενή συνεργασία με όλους σας. Ευχαριστώ. Η επόμενη συζήτηση τώρα ε, μάλλον επί του θέματος αυτός η επόμενη συζήτηση θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου. Ε, τώρα θέλω να σας πω ότι η προθεσμία για τροπολογίες για την έκθεση του κυρίου Σούστας για τις προκηρύξεις δημοσίων προμηθειών ε, είναι για τις 17 Ιουλίου 6 το απόγευμα και όσον αφορά ε, την ε, έκθεση για τον κανονισμό για, τις για την οδηγία για τις παραχωρήσεις θα παραμείνει ανοιχτό δεν ξέρουμε ακόμη αν θα λάβουμε απόφαση και θα αποφασίσουμε το Σεπτέμβριο τώρα χαιρετίζω τους εκπροσώπους του ε, Διεθνού Οργανισμού ε, Εργασίας ε, με τους οποίους θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεως, απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ ο, ο ε, επικεφαλής Γενικής Διευθύνσεως και ο κύριος Ρούντι Ντελάκα, εκπρόσωπος του Γραφείου των Βρυξελών και τους δίδω τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά σήμερα ήρθα εδώ για να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή των απόψεων και των ε, πληροφοριών όσον αφορά κάποιε χώρε που σας ενδιαφέρουν. Ο, το Διεθνέ Γραφείο Εργασία. Ε, εκτιμά την ευκαιρία που δίνεται για συνεργασία με διάφορα θεσμικά όργανα στην Ευρώπη, ούτω ώστε να μπορούμε να προωθήσουμε αυτό που θέλουμε πάντα στον κόσμο. Και από ό,τι γνωρίζω, οι ανταλλαγέ μα απόψεων τώρα, εν ώψη αυτών των νέων συμφωνιών, ε, ε, έχουν γίνει πιο πυκνές, ούτω ώστε μπορούμε, έτσι μπορούμε να προωθήσουμε αυτά τα πρότυπα, τα στάντα εργασία που θέλουμε και εμεί και εσείς και αυτό γίνεται ε, μια από την, την θα έχουμε την ανθεώρηση του στιγμούς Γενικευμένων Προτιμήσεων και προσπαθούμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με ε, κάποιο είδους ε, διαδικασία καινούργια όσον αφορά την διαχείριση κάποιων καταγγελιών και έχουμε επίσης και κάποιους ανεξαρτήτους εμπειρογνώμονες και τριμερή όργανα. Οπότε οι αποφάσεις αυτών είναι σημείο αναφοράς όσον αφορά το, το, το, το πώς θα υπάρχει αξιοπρεπής εργασία για όλους. Σε σχέση με αυτό, επομένως, ε, συμφωνούμε με τους στόχους σας, με τις πολιτικές αξιολογήσεις, ε, πάνω σε αυτήν ε, την, την, την, την, την, Επιτροπή των Εξαρτήτων Ειδικών σε αυτές τις δύσκολες ώρες και σε σχέση και με τα τριμερή μας φόρα. Οπότε γι' αυτό και θα πρέπει να πούμε πόσο σημαντικό είναι το ότι έχουμε πρόοδο σε διάφορα μέτωπα όπου βέβαια ακόμα επιδέχεται βελτίωση η κατάσταση και γι' αυτό χρειάζεται να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τα πράγματα ε, στον πραγματικό κόσμο, οπότε θέλουμε να δούμε τώρα πώς θα έχουμε βελτίωση των προτύπων εργασίας σε διάφορες χώρες και προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε βήματα πρώτα. Οπότε η συμφωνία αυτή να μπορεί με την Κολομβία, είναι πολύ σημαντική και εκεί επομένως και στο δίκαιο στο δημοτικό θα βελτιθεί κατάσταση με αυτή τη συμφωνία και οι υποπτικές αρχές ε, είπαν ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα όσον αφορά τη συμφωνία της σύνδεσης. Έχουμε μια έκθεση της ε, αποστολής της Τριμερού το 2009 και είπαν πόσο σημαντικό είναι να αναβαθμιστεί ο κοινωνικό διάλογος, να ληφθούν κάποια μέτρα κατά της ατιμορρησίας, κατά της βίας, να αρθούν κάποιοι φραγμοί όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, ε, για να γίνουν κάποιες ε, επιθεωρήσεις στην εργασία, να έχουμε μόνο σε τέτοιους από αυτή την ειδική επιτροπή ε, για τις καταγγελίες όπου κρυμούσαν κάποιες καταγγελίες και τις διεκπαιριώσαμε. Θέλουμε επίσης να υπάρχει ειδική εκπαίδευση κάποιων εισαγγελέων, γενικά διοικητικών οργάνων και δικαστικών για τα δισεκατοντάδες των, ε, των, των επεισοδίων ει βάρος συνδικαλιστών. Πάντως οι πολιτικές αρχές συνεχίζουν να καταδικάζουν τους φόνους ε, των ε, συνδικαλιστών και την άσκηση βία γενικά Οπότε, να ανέψει δράση χρειάζεται συνεργασία με τις ΗΠΑ και έτσι να δυναμώσουμε ε, το, το, το κράτος ε, της ε, Κολομβίας και να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα ιδίω ιδίως όσον αφορά την, την, το, το και τα δικαιώματα εργαζομένων. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο να δούμε τι θα γίνει με κάποια προστατευτικά μέτρα, κάποιες καμπάνιες προφοριακές, κατάρτιση επομένως δικαστών, αστυνομικών κλπ ε, ούτω ώστε να σταματήσουν αυτά τα βία εγκλήματα που γίνονται και έτσι να υπάρχουν ε, ε, αυθεντικές συλλογικές συμβάσεις ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς θα υπάρχει πάλι μία, μία διαμεσολάβηση πώς θα υπάρχουν όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για την εργασιακή αγορά και επίσης Γενικότερα στη Λατινική Αμερική πολλές φορές υπάρχει το πρόβλημα το ότι δεν υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί κρατικοί. Ε, δεν υπάρχει ονικό διάλογος. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε διάφορες χώρες στην περιοχή αυτή οι οποίες έχουν ε, μιμηθεί την Κολομβία για τη βοήθεια του ILO εκεί ούτω ώστε να υπάρχει διαμεσολάβηση, να υπάρχει ε, κάποιο είδου ε, επίλυση των εργασιακών διαφορών. Φιλιππίνες. Εκεί είδαμε τι γίνεται όσον αφορά τα όσα γίνονται από τους εμπειρογνώμονες, τι, γίνεται από αυτές τις τριμερείς επιτροπές όσον αφορά την ελευθερία του συντελείστα και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε μια αναβαθμισμένη συνεργασία και επίσης όσον αφορά το πρόγραμμά μας για την ελευθερία του συντελέστα οι κατευθυντέ γραμμέ και η όλη συμπεριφορά των διαφόρων Υπουργείων Εργασία Εσωτερικών, Αμήνη, δικαιοσύνη, ένοπλε δυνάμει ε, και στην κοινωνία των Φιλιππίνων όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων και των δραστηριοτήτων και η πρώτη απόφαση που είναι σημαντική και κάνει διάκριση μεταξύ ε, της δραστηριότητα ενός ε, μέρους συνδικάτου και τη δολοφονία του και αναφέρεται ότι θα τιμωρούνται από τούτο και στο εξή πολύ σοβαρά. Λοιπόν, και έχουμε επηρεάσει και τα καταναγκαστική εργασία στο Μιανμάρ ε, μετά από πολλές επικρίσεις ψηρά ετών που συνδυαζόταν με επικοδομητικέ δεσμεύσεις για βελτιώσει και προσπάθειες βελτιώσει. Όπως γνωρίζετε, η Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας ε, δέχτηκε τα τίματα των μελών όσον αφορά τι εμπορικές σχέσεις με το Μιανμάρ και την επιβολή κυρώσεων και αναφερόμαστε στο, στην αναθεώρηση προτεραιοτήτων δράσεων για την εξάλληψη όλων μορφών υποχρεωτική καταναγκαστική εργασία, καθώ και τι πρόοδο συνέβη, ώστε να υπάρχει η πλήρη ε, ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Ε, και υπάρχει ειδική ομάδα στη Γιανγκόν πάνω σε αυτό το θέμα. Εποπτικοί φορεί επί μακρόν σχολίαζαν την ανάγκη η κυβέρνηση του Πακιστάν να αλλάξει την νομοθεσία τη, ούτω ώστε να συνάδει με τι βασικέ προδιαγραφέ για την εργασία. Το 2010 αναφέρθηκαν ανησυχίε όταν υπήρξαν προβλήματα σε επαρχίε με εργασιακά θέματα και υπήρχε νομικό και ενό αφορά το κοινωνικό διάλογο και το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε. Οι τριμερεί ε, επαφές οδήγησαν σε νέες διευθετήσεις όσον αφορά τις ε, σχέσεις της εργασιακές της πρωτεύουσας πρωτεύουσας, αλλά υπήρχαν διαφορές μεταξύ του νόμου και των συμβάσεων. Δυστυχώς, οι υποπτικοί μηχανισμοί είδαν ότι αύξησε και αυξήθηκε και η παιδική εργασία λόγω αύξησης της φτώχειας. Η νομοθεσία απαγορεύει τα παιδιά να συμμετέχουν σε συγκρούσεις και εχθροπραξίες, αλλά όλο και περισσότερο γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούν τα παιδιά για ενόπλες σειράξεις και στην ταπιτουργία χρησιμοποιούνται πολλά παιδιά στην εργασία και εκφράσαμε έντονες ανησυχίες για τον αριθμό των παιδιών, των ανηλίκων που δεν πηγαίνουν σχολεία με πολύ μικρή ηλικία. Και δεν εφαρμόζουν σωστά οι νόμοι για την απαγόρευση τη παιδική εργασία, διότι δεν γίνονται αρκετέ επιθεωρήσει. Το Διεθνέ Πρόγραμμα για την Κατάργηση Εργασία των Παιδιών, IPEC, έχει ένα πρόγραμμα επιτόπου, χρηματοδοτείται αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να υπάρξουν μονάδε σε ομοσπονδιακό και επαρχιακό επίπεδο, μονάδε που θα ελέγχουν κατά πόσο εφαρμόζονται τα προγράμματα, τα διεθνή για την εξάλληψη τη παιδική εργασία και την αποκατάσταση των παιδιών εργατών. Λοιπόν, στη Γεωργία πρέπει να γίνουν προσπάθειες να αλλάξει το εργασιακό δίκαιο για να συμμορφωθούν με το δικαίωμα της συντερίζεστε δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις αλλαγές η κυβέρνηση. Έγιναν δύο αλλαγές. Το ILO βοηθούσε την κυβέρνηση κοινωνικού εταίρους να δημιουργήσουν μηχανισμό διαμεσολάβηση, ώστε πιο γρήγορα να αντιμετωπίζονται προβλήματα από ότι υπάρχουν παραβιάσει ε, δικαιωμάτων των συνδικάτων όσον αφορά την εργασία των παιδιών. Οι υποπτικοί φορεί δήλωσαν ότι υπάρχει σχέδιο δράση για την καταπολέμηση του εμπορίου παιδιών για το 2009-2010 αλλά παρατήρησαν με τα ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας έχουν καταργηθεί και αυτό αποδεινόμενο τις σχετικές δράσεις για την μείωση της εργασίας, την κατάργηση της εργασίας των παιδιών, κάτι και όταν γέννη. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστεί το εφαρμογή του κράτους δικαιώματα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν ε, προσπαθήσει να εφαρμόσουν τις βασικές ε, συνθήκες για τη σωστή εργασία. Λοιπόν, οι φορείς επιθεώρησης μπορούν να βοηθήσουν να μην τα δικαιώματα. Ο επιθεωρητικό φορέα μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, να συλλέξει στοιχεία, να βοηθήσει τον εντοπισμό ιδιαίτερα βαλωτήτων τομέων ή ομάδων και να επεξεργαστούν τα διάφορα ιδιωτικά μέτρα. Οι υποπτικοί φορεί λοιπόν τονίζουν ε, την υποστήριξη των επιθεωρήσεων οικονομικά με ανθρώπινου πόρου και κατάρτιση όσον αφορά τι διεθνεί πρωτογραφέ. Οι υποπτικοί φορεί παρακολουθούν με τα ανησυχία στη χρήση τη εργασία των παιδιών σε κάποιου τομεί όπω είναι ο βάμβαξ και η παραγωγή ε, ε, κακάου. Και έγιναν σχόλια όσον αφορά το Ζερμπαϊζάν, την Κίνα, το Καζακστάν, Κυργιστάν, Τατζικιστάν αλλά και ο Ουσμπεκιστάν. Σε περισσότερε περιπτώσει η χρήση των παιδιών για το μάζεμα βαμβακίου απαγορεύεται δια νόμου, αλλά δεν εφαρμόζεται. Η IPEC έδινε τεχνική αρρωγή σε κάποιες χώρες Κεντρικής Ασίας από το 2005. Το Σμπεκιστάν συζητήθηκε ιδιαίτερα από τους επαπτικούς μηχανισμούς και λήφθησαν διάφορες αποφάσεις της τριμερούς επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των προδιαγραφών. Και το Διεθνές Συνδικαστικό Κίνημα και οργανώσεις εργοδοτών είδαν να χρησιμοποιούνται πολλά παιδιά κατά τη συγκομιδή του βάμβακος αλλά υπάρχει και κινητοποίηση από πλευρά κρατών σε κάποιες περιπτώσεις. Η υπηρεσία μας συζητά με την κυβέρνηση πρόσφατα, συζήτησε, όμως δεν δέχτηκε όμως την πρόσκληση για τριμερείς αποστολές εποπτείας η κυβέρνηση. Ούτε κάλεσε αποστολή μας για να κάνει εξολόγηση της κατάστασης όσον αφορά ε, τη χρήση παιδιών για τη συλλογή βάμβακος. Και στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας δεν συζητήθηκε το θέμα. Θεωρήθηκε σημαντικό να αναθεωρηθεί η εφαρμογή της σύμβασης φέτος. Θέλαμε νέα κυβερνητική έκθεση για να εξεταστεί από του εμπειρογνώμονε. Στην επόμενη συνεδρίαση θα γίνει Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Και για άλλε χώρε ισχύει αυτό. Λευκορωσία, Κολομβία, Γουατεμάλα, όπου ζητήθηκε επιτροπή έρευνα, Μιανμάρ επίση, Πακιστάν. Η εργασία των παιδιών στην παραγωγή κακάου ε, υπάρχει στην Κάνα και ακτή ελεφοντεστού. Το IPEC πιστεύει ότι 1,7 παιδιά, 1,7 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται. Η ακτή ελεφαντοστού είπε ότι θα ερευνήσει στα πλαίσια του σχεδιου δρασεω δράσεως 2007-2009 το είχε πει, είχε υποσχεθεί. Η Γκάνα εφάρμοσε εθνικό πρόγραμμα ε, από το 2006. Η Γκάνα μέσω του προγράμματος άρχισε ευαισθητοποίηση για το θέμα ξεκίνησε και ένα πρόγραμμα υποστήριξη διαβίωση για να αυξήσει το έσοδο των εργαζομένων στον τομέα του κακάου και να μπορέσει να βοηθήσει μέσω κυβερνητικών μηχανισμών τα παιδιά να επιστρέψουν στα σχολεία. Το ΑΕΛΟ κινείται και με συμπράξει ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ώστε να εξαλειφθεί η εργασία των παιδιών στον τομέα παραγωγή κακάου στην Αφρική. Είναι σημαντική η ελευθερία του συνεταιρίζεστε είναι δικαίωμα για να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό προωθούμε την ελευθερία του συντερίζεστε και στι απομακρυσμένε περιοχέ τη Υπέθρου. Ευαισθητοποιούνται οι εργαζόμενοι για τα δικαιώματά του, για την καταπολέμηση τη καταναγκαστική εργασία και την εργασία των παιδιών. Η ελευθερία του συνεταιρίζεστε σχετίζεται με τη δράση των διαφόρων φορέων, κυρίω στην Υπέθρο, για την εξάλληψη τη εργασία των παιδιών. Ελπίζω αυτά που σας είπα να ήταν χρήσιμα και προσβλέπω σε τυχόν σχολιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Ήταν πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλοί αριθμοί και θα ήθελα να μας δώσετε την ομιλία σας κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να την μοιράσουμε. Έχω τέσσερις ε, υποψηφίους που ζητούν το λόγο και πρώτος είναι ο κύριος Κούτας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή είμαι ο εισηγητής για το πρωτόκολλο των ε, ε, κλωστεφαντουρχικών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Ουσμπεκιστάν έχω ορισμένα ερωτήματα. Καταρχήν, υπάρχει μία πραγματική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ουσμπεκιστάν για την αποδοχή της αποστολής της τεχνικής βοηθείας 2012-2013 ε, ε, ε, τι πιστεύετε υπάρχει περίπτωση να δεχθεί το Ουσβεκιστάν μέχρι τέλος Ιουλίου που είναι η προθεσμία που έχετε καθορίσει Επίσης γνωρίζετε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάτι παραπάνω για να βοηθήσει το διάλογο μεταξύ ε, της ε, κυβερνήσεως του Ουσμπεκιστάν και της Ευρωπαϊκής της για να γίνει δεκτή η αποστολή διότι την τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει την εργασία των παιδιών στο Ουσμπεκιστάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε εξηγήσει ότι Υπάρχει μία τριμερής επιτροπής ε, ε, η οποία συνεδριάζει στην ε, Γενέβη και δεν έχει εστιαστεί συγκεκριμένα στο Ουσμπεκιστάν. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, δεν ενδιαφέρεται πλέον ο οργανισμός σας για τα παράπονα σχετικά με το θέμα αυτό. Επίσης αναφέρατε διάφορες χώρες όπου πιστεύετε ότι τα δικαιώματα των παιδιών παραβιάζονται. Θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε ένα κατάλογο των χωρών αυτών πέραν του Ουσμπεκιστάν όπου παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών. Με ενδιαφέρει να δω τι μπορείτε να μας δώσετε και τέλος αναφέρομαι στους λίγους εκπροσώπους ε, της ε, συναδέλφους της Επιτροπής που είναι ακόμη εδώ και να τους ρωτήσω εάν πιστεύουν σε περίπτωση που η κυβέρνηση του Ουσβεκιστάν δεν δεχθεί ε, την αποστολή η οποία έχει ε, υιοθετηθεί στην Ολομέλεια και στην ενδιάμεση έκθεση, τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να υπάρξει μία άλλη περίοδος συγκομιδής και να δούμε αν ε, οι Ουσμπέκοι θα δεχθούν του χρόνου μία εκπροσώπηση και αποστολή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και θα πρέπει να κατατίσουμε ένα καλό πρόγραμμα για να δούμε πώς θα, δεν θα συνενέσουμε στο πρωτόκολλο αυτό. Είναι μία πρόταση που διατυπώνω και σας παρακαλώ να συμφωνήσετε μαζί μου να βρούμε την καλύτερη λύση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό και ζητώ από ε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας να κοιτάξει τι γίνεται με τη συγκομιδή. Ο κύριος Μάρφη. Έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν ε, για το Ουσμπεκιστάν, ε, όπως είπε και ο Φραλαλής σας αντιλήφθηκα ότι υπάρχουν ε, διαπραγματεύσεις για μια τεχνική αποστολή στο Ουσμπεκιστάν. Αν ναι, μπορείτε να μου δώσετε ορισμένες λεπτομέρειες, δηλαδή πότε θα μεταβεί η Επιτροπή που θα ήταν καλό να γίνει αυτό στο τέλος της εποχής συγκομιδής και εάν είναι μία αποστολή τεχνικής βοηθείας ε, πώς ε, θα αναγνωριστεί ε, στα πλαίσια αυτά ο ιδιάζων λόγος της κοινωνίας των πολιτών. Επίσης το θέμα της, της χρήσεως παιδιών την καλλιέργεια του βάμβακα πέραν της συγκομιδής κατά την σπορά παραδείγματος χάρη. Τι γίνεται, δεν έχω ακούσει τίποτα και τρίτον, στο Καζαστάν, μήπως μπορείτε να μας πείτε εάν υπάρχει μια, κάποια δουλειά που κάνετε εκεί διότι φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική υποχώρηση ε, υπάρχει γενοκτονία, ε, μία υποβάθμιση των δικαιωμάτων των πολιτών και θα ήθελα να ξέρω αν γνωρίζετε ότι έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει η νομοθεσία στις 17 Φεβρουαρίου εφέτος και ε, εμποδίζει την, ε, το δικαίωμα ελεύθερης ε, συνέλευσης, μειώνει τα δικαιώματα των εγγύων γυναικών που εργάζονται, μειώνει τις δυνατότητες προσφυγής στις διαπραγματεύσεις απολύσεως και ούτω καθεξής. Ε, σχετικά με την ε, Κολομβία που μας ενημερώσατε για ορισμένα θέματα. Γνωρίζετε τι γίνεται σχετικά με τον καθορισμό ενός ανωτάτου χρόνου εργασίας. Ευχαριστώ κύριος Ντάρμουθ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω την εξαιρετική εργασία που έκανε ο, η, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας για να καταπολεμήσει την εργασία των παιδιών. Και θα ήθελα να ρωτήσω το γραφείο σας ε, ε, ε, κάτι συγκεκριμένο το οποίο κυκλοφόρησε στις αγγλικές εφημερίδες και σε γενικές γραμμές σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ μία, ένα ισπανικό, μια ισπανική συνδικαλιστική οργάνωση παρέπεμψε την περίπτωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν θυμάμαι, ότι ε, αν ένα παιδί ε, αρρωστήσει ε, εις, της, κατά τη τις ε, αργίες προστίθεται ο χρόνος ασθενείας ή στις αργίες. Όπως ξέρετε στη χώρα αυτή υπάρχει 25% περίπου ο χρόνος αδείας. Λέγεται όμως ότι ε, ενώ ένας ε, τέτοιος κανονισμός σχετικά με την εργασία ε, μπορεί να ισχύσει ε, εμποδίζει και αποτρέπει τους εργοδότες από το να προβούν σε προσλήψεις. Εμείς λοιπόν είμαστε αντίθετοι στην πολιτική μας ομάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να καταρτίζει ε, εργατική νομοθεσία για το Ηνωμένο Βασίλειο ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος της ερωτήσεώς μου. Ήθελα να ξέρω εάν ε, η για οποιαδηποτε αλλη χωρα αλλα δεν ειναι αυτος ο στοχος τη ερωτησεω μου ηθελα να ξερω εαν η οργανωση σα στήριξε ε, την προσφυγή της, του, της Ισπανικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και επανερχόμενος στη δήλωση που έκανα προηγουμένως ότι αυτό μπορεί να αποτρέψει ε, τους ε, εργοδότες να ε, προσλαμβάνουν σε μια εποχή τεράστιας ανεργίας στην Ισπανία. Πιστεύετε ότι κατά τη γνώμη σας αυτή η άποψη είναι εγκυρή ε, ε, δηλαδή ε, έχει κάνει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας κάποια έρευνα σχετικά με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να είναι πολύ σύντομες οι ερωτήσεις γιατί έχουμε 10 το πολύ 15 λεπτά. Ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη παρουσίαση και από την πλευρά μου θα ήθελα να ξέρω κάποια πράγματα παραπάνω όσον αφορά τις λεπτομέρειες των προσπαθειών που κάνετε έναντι του Σμπεκιστάν. πότε θα υπάρξει επιτόπια αποστολή τι γίνεται όσον αφορά με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών ε, και μη κυβερνητικέ οργανώσεις που θα μπορούσατε επιτόπου να συναντήσετε. Οι ουσμπεκικές αρχές τι λένε. Τι σας λένε. Αρνούνται την ύπαρξη του προβλέματος. Θεωρούν ότι το επεξεργάζονται το θέμα και χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω. Θεωρούν ότι είναι κάτι που εφευρίσκουν τα διεθνή ΜΜΕ, διεθνείς οργανισμοί. Πώς δικαιολογούν αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Δεύτερον, για το Σμπεκιστάν. Βάσει και των όσων είπε ο κύριος Κούτας. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να βιαστούμε να πάμε στην Ολομέλεια. Όσο εκρεμεί η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, έχουμε περιθώριο για ελιγμούς, για διαπραγματεύσεις. Και ίσω ελπίζω για επιτόπιε βελτιώσει. Από τη στιγμή που θα γίνει η ψηφοφορία και είναι αρνητική η ψήφο, κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε καμία επιρροή πια ή τουλάχιστον πολύ μικρότερη όσον αφορά τα τεκτενόμενα στο Σμπεκιστάν. Εγώ θα το πρόσεχα αυτό. Ήδη είναι η κατάσταση ε, που φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση του Σμπεκιστάν ότι υπήρχε τη ψηφοφορία και ότι δεν συμφωνούμε και συζητάμε. Έχουμε ελάχιστο χρόνο, αλλά μπορείτε να μας πείτε κάτι για την εργασία των παιδιών στην Ινδία Εγώ είμαι συγκεκριτής και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το βασικό πρόβλημα για την ώρα συνομιλίε με την Ινδία. Δύσκολο να πουλήσουμε αυτή τη θέση προ τους Ινδούς ομολόγους μας. Θα ήταν ευπρόσδεκτη τυχόν πρότασή σα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να προσθέσω δύο ερωτήσει. Πρώτον, θα ξέρετε ίσως το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα για την Κολομβία και το Περού. Ζητήσαμε έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργατικών δικαιωμάτων και φαίνεται ότι είναι πρόθυμη η κυβέρνηση της Κολομβίας να παρουσιάσει ένα τέτοιο δικό χάρτη. Θα μπορούσε ο ΑΕΛΟ να βοηθήσει την παρακολούθηση της εφαρμογής τέτοιου δικού χάρτη. Δεύτερον, εδώ και ένα χρόνο ε, έχει τεθεί σε ισχύ η συμφωνία με την Νότια Κορέα Υπάρχουν κάποιες απαιτήσει από την πλευρά μας όσον αφορά τις βασικές, τα βασικά εργατικά δικαιώματα. Ξέρετε τι γίνεται όσον αφορά τα προβλήματα για τα προβλήματα των εργαζομένων. Βελτιώθηκε η κατάσταση λόγω της εμπορικής συμφωνίας και των εμπεριεχομένων απαιτήσεων που επιβάλαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να σχολιάσει. Η κυρία Σάντο, ευχαριστώ που δίνει το λόγο. Για το Ουσμπεκιστάν, έχω μια ερώτηση και έτσι κλείνει το μικρόφωνο. Ξανακλείνει το μικρόφωνο. Δεν ακούσαμε την ερώτηση. Α, τώρα είμαστε συνδεδεμένοι. Επιβεβαιώνω ότι επανειλημμένα στο διάλογό μας με το Ουσμπεκιστάν στηρίξαν θέση του ILO και να βοηθηθεί στην εποπτεία. Βασικό αυτό για την Κορέα. Θα σας δώσουμε πρόσφατες πληροφορίες. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν συναντήσεις. για το κεφάλαιο περιβιωσιμότητας. Πήγαν πολύ καλά οι συνομιλίες. Καλά ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις. Τι είπατε... Για το ισπανικό θέμα θα δώσω το λόγο στη Γενική Διεύθυνση την υπεύθυνη για την απασχόληση. Νομίζω τα κάλυψα όλα. Θυμήστε να ξέχασα κάτι. Εν γέννη, για τα θέματα GSP, παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τι γίνεται από πλευράς ελέγχου, κατά πόσο πρέπει να παρέμβουμε όσον αφορά το γενικό σύστημα προτιμήσεων, πώς εφαρμόζονται οι προδιαγραφές κλπ. Ευχαριστώ Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Λοιπόν, μία σύντομη παρατήρηση ε, σχετικά με τον χρόνο εργασίας ε, στην Ισπανία είναι μια ε, ρύθμιση που διέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, και ε, δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να θυγεί στα πλαίσια των εμπορικών, ε, των εμπορικών σχέσεων. Ο κύριος Ντάρτμουθ, τα μέλη της Επιτροπής θα αποφασίζουν τι θέματα θα φύγουν. Αν σέβεστε την Επιτροπή, πρέπει να μας σέβεστε. Έχουμε δει αυτό το ερώτημα στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας και έθεσα ένα θέμα που απασχολεί τους ψηφοφόρους μου. Ε, θεωρώ ότι η απάντησή σας δεν είναι ούτε ικανοποιητική ούτε σέβεται την Επιτροπή εάν δεν μπορείτε να μου απαντήσετε τώρα θα σας παρακαλούσα να μου απαντήσετε γραπτός και απευθύνω την παράκληση αυτή μέσω ο, της Προεδρίας ε, το λόγο έχει τώρα το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Τα γενικά σχόλια που έχω να κάνω θα τα παρουσιάσω και μετά θα δώσω το λόγο στη συνάδελφό μου η οποία έχει ασχοληθεί με αυτές τις διαπραγματεύσεις του Μπακιστάν για την αποστολή και θα σας ενημερώσει. Καταρχήν όμως επαναλαμβάνω και πάλι ότι το γεγονός ότι το Ουσμπεκιστάν δεν έχει συζητηθεί φέτος στην Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας δεν έχει καμία σχέση με την ε, εφαρμογή της ε, Σύμβασης Εργασίας στο Ουσμπεκιστάν. Ε, ε, δεν είναι ε, αποτέλεσμα ότι το, του γεγονότος ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Εργασίας λέγει ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε πλέον με το Ουσμπεκιστάν. Όλοι μαζί ζήτησαν να παρακολουθήσουμε την πορεία, να επανέλθουμε και του χρόνου ή στη διάσκεψη θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τη συζήτηση αυτή. Όσον αφορά την παρακολούθηση του χάρτη πορείας στην Κολομβία, έχουμε εμπλακεί, έχουμε δώσει πληροφορίες ε, για τον χάρτη πορείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό, διότι τώρα ξεκινάμε το φθινόπωρο αυτή την εργασία στην Κολομβία ιδίω όσον αφορά την ε, ελευθερία του συνέρχεστε ε, και ουσιαστικά θα το παρακολουθήσουμε για την επόμενη τριετία και θα σας ενημερώνουμε. Νότιος Κορέα. Μας ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης ε, θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω ε, οι κοινωνικοί επέροι έχουν εμπλακεί στη συζήτηση αυτή διότι την τελευταία φορά που πήγαμε στην Κορέα Νότιο Κορέα δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία οι κοινωνικοί εταίροι ήθελε ε, να δεν ήθελαν να ασχοληθούν με την πτυχή των προδιαγραφών εργασίας της συμφωνίας και αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια όχι μόνο στην τελευταία και πρόσφατη σύμβαση εργασίας αλλά και στην πρώτη και όσον αφορά την ελευθερία του συνέχεια ε, είναι κάτι το οποίο η αρμόδια επιτροπή παρακολουθεί. Και τώρα, ε, χωρίς να έχουμε ξεχάσει την ερώτηση ε, των Ισπανών, θα πανέλθουμε, θα δώσω λόγο στην συνάδελφό μου. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Πολλές ερωτήσεις ετέθησαν, αλλά βασικά οποιαδήποτε πραγματική πρόοδος όσον αφορά την τεχνική επιτόπια αποστολή είναι το θέμα. Μετά από τις δύο συμβάσεις ζητήθηκε από την κυβέρνηση να δεχτεί μια επίσκεψη τριμερών παρατηρητών και ήταν σαφές ότι δεν το δεχόταν αυτό. Το Φεβρουάριο του 2012 ίσως λόγω βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από ό,τι μου είπαν Μα είπαν ότι θα καλούσαν το Διεθνέ Γραφείο Εργασία για μια τεχνική συμβουλευτική επιτροπή τον Μάιο 2012 στα Σκένδη. Πήγε η υπηρεσία, πήγα κι εγώ. Ήταν παρούσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτόπου και κατά τη διάρκεια τη αποστολή ήταν σαφέ ότι δεν δεχόταν υψηλού επίπεδου τριμερή αποστολή εποπτεία αλλά θα δεχόταν μια αποστολή του διεθνού Γραφείου Εργασία. Ε, και παρακολούθηση από την ΆΕΠΕΚ σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Το είπαν αυτό το Μάιο διότι τους είπαν ότι πιθανότατα θα συζητηθούν αυτά τον Ιούνιο στη διάσκεψη. Η... Το συμπέρασμα ποιο ήταν. Από ό,τι μας είπαν θα δεχόταν μία αποστολή του γραφείου που θα, το ακολουθούσε ένα εργαστήριο το τριμερές. Υπήρξε συνάντηση πέντε φορές με την ε, τριμερή αντιπροσωπεία του Ουσμπεκιστάν. Στην αρχή δήλωσαν κάποια προθυμία να καλέσουν το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για μια τέτοια αποστολή. Προς το τέλος της διάσκεψης όμως είπαν τεχνική βοήθεια για αυτούς σημαίνει πολλά περισσότερα δημιουργία δυναμικού, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση ε, και εκπαίδευση των υπευθύνων για την επιθεώρηση εργασία και ότι είχαν πάρα πολύ καλό σύστημα εποπτείας υπό τη μορφή ε, ομάδας εργασίας ε, της αρμόδιας διεύθυνσης και εμεί είπαμε ότι μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά και να του βοηθήσουμε και με την νομοθεσία. Αλλά εποπτεία θα ήταν συνιστόσα. Δεν συζητήθηκε το θέμα τον Ιούνιο. Αυτό μας είπαν ότι δεν τους είπαν ότι δεν θα ξέφευγαν από τον έλεγχο γιατί η ομάδα εμπειρογνωμόνων τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα εξακολουθούσε να εξετάζει την υπόθεση. Τέλος Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, μας είπαν ότι μέσα Ιουλίου θα επέστρεφαν, θα απευθυνόταν ξανά προς το γραφείο, εξακολουθούν οι διαπραγματεύσεις, θα τους συναντήσουμε. Λοιπόν, μέσα Ιουλίου θέλαμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της Τεχνικής Επιτροπής εποπτείας. Η αποστολή αυτή θα έχει πλήρη πρόσβαση. Ε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς τα που το πάνε. Ακόμα συζητάμε πότε θα γίνει η αποστολή. Η υπηρεσία συναντήθηκε με την UNICEF. Το γραφείο με τη συναντήθηκε με την UNICEF. Πήγε στην Τασκένθη η UNICEF, συναντήθηκε με προσώπου του, γραφείου, της, του Υπουργείου Εργασία και είναι πολύ απεσιόδοξη η UNICEF. Ήδη φυτεύτηκαν οι σπόροι του βάμβακος φέτος ένα μήνα νωρίτερα. Άρα και η συγκομιδή του βάμβακος θα γίνει ένα μήνα νωρίτερα. Άρα, αν κάνα μια αποστολή, θα έπρεπε να γίνει ακόμα νωρίτερα. Και το θέμα των θεωρήσεων είναι πολύ χρονοβόρο. Τον... Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, κάνουμε κάθε προσπάθεια, όμως αυτά. Άλλη ερώτηση. Τι λέει η κυβέρνηση για όλα αυτά ήταν η ερώτηση. Λένε ότι δεν δέχονται όλα αυτά. Ότι έχουν, έχουν 100% αλφαβητισμό. Όλα τα, όλα τα παιδιά ξέρουν γράμματα. Πάνω όλα τα παιδιά στο σχολείο. Είδαμε τον Υπουργό Υγεία και τον Υπουργό Παιδεία. Είπαν τελευταία 20 ετία είχαμε πάρα πολύ σημαντική πρόοδο σε αυτό το θέμα. Δεν δέχτηκαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει έχουν δικό του σύστημα εποπτείας. Και κάποιος είπε, θεωρούν ότι είναι στόχος. Ναι, θεωρούν ότι είναι στόχος κάποιων ε, τομέων της διεθνούς ε, κοινότητας. Αυτά έχω να σας πω. Uh, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν νομίζω ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα και όλες τις ερωτήσεις. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε πλέον χρόνο. Ενδεχομένως μπορείτε να κάνετε ορισμένες διμερείς συζητήσεις και διμερείς ανταλλαγές πληροφοριών. Ελπίζω να έχετε καλές διακοπές κατά το καλοκαίρι, να φρεσκάρετε το μυαλό σας και θα ξαναβρεθούμε στις 3 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ.